Prego prendere posto. Παρακαλώ καθίστε. Θα ξεκινήσουμε με μια κάποια καθυστέρηση είναι αλήθεια. Υπήρξε μια ταξία και χθε και σήμερα το πρωί με τα αεροπορικά δρομολόγια και κάποιοι από τους συμμετέχοντες βουλευτές από τα κοινοβούλια θα έλθουν μένα αλλά με καθυστέρηση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίαση καλύπτεται τηλεοπτικά και αναμεταδίδεται ε, στο διαδίκτυο. Να ευχαριστήσω όλος ιδιαιτέρως τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων Δεκαεννέα χώρες συμμετέχουν ή θα συμμετέχουν στη συνάντησή μας ίσως 18. Ξέρετε ότι έχουμε ψήφο εμπιστοσύνης στη Γερουσία α, για την κυβέρνηση Μπερλουσκόνη και αυτό θα προκαλέσει καθυστερήσεις στους Ιταλούς βουλευτές. Αλλά παρόλα αυτά 18 χώρες είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για την παρουσία σας. Όπως γνωρίζετε το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λισαβόνας καθορίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα στενό συντονισμός ανάμεσα στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα θεσμικά όργανα. Με στόχο μια πιο γρήγορη και αποτελεσματική ε, πορεία ολοκλήρωσης. Θα συζητήσουμε θέματα λοιπόν που μας ενδιαφέρουν, θέματα κοινού ενδιαφέροντος, οι συζητήσεις αυτές δεν θα πρέπει να γίνονται μόνο σε σύνολο των, σε επίπεδο συνολικά των κοινοβουλίων, αλλά και σε επίπεδο των ε, μεμονωμένων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Και έτσι θα δοθεί η δυνατότητα και στους βουλευτές των κρατών μελών να λειτουργήσουν ελεγκτικά και να λειτουργήσουν και σαν μια επιπλέον όθηση προς τις κυβερνήσεις τους, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε μια ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ουσιαστική. Δύο θέματα θα έχουμε σήμερα για συζήτηση. Πολύ σημαντικά. Τώρα το πρωί θα μιλήσουμε για την ενιαία εκλογική διαδικασία, την προοπτική της ενιαίας εκλογικής διαδικασίας. Είναι ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τα κράτη-μέλη και ανεξάρτητα από το ποια θα είναι απόφαση που θα ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο θα κληθεί να επικυρώσει την πιθανή τροποποίηση της συνθήκης της πράξης ε, του 1976 σχετικά και με το καθεστώς των Ευρωβουλευτών και κυρίως σχετικά με τις διαδικασίες εκλογής τους. Το απόγευμα θα συζητήσουμε για μια καινοτομία η οποία θα έλεγα είναι από τις πιο χαρακτηριστικές ε, της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, την λεγόμενη πρωτοβουλία των πολιτών. Ξέρετε ότι ένα εκατομμύριο πολίτες που θα πρέπει να ανήκουν σε ένα σημαντικό αριθμό μελών μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκινήσει την νομοθετική διαδικασία μια συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών είναι να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στον πολίτη. Ήδη είχαμε εκθέσεις από 12 χώρες προ την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε τη συζήτηση Η συζήτηση και για τον ενιαία εκλογική διαδικασία και για την πρωτοβουλία των πολιτών εμείς απλά να πάρουμε αποφάσεις, αλλά θα πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να συλλέξουμε τις τροπολογίες και τροποποιήσεις που θα προτείνουν οι συνάδελφοι και να καταλήξουμε σε χρήσιμες συστάσεις. Έχετε ήδη λάβει το πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, της σημερινής μέρας συνετάχθη το πρόγραμμα αυτό και ε, μετά από συνεννοήσεις με τα κοινοβούλια των κρατών μελών ελπίζω να σας ικανοποιεί το πρόγραμμα και να μην προκαλεί κάποια δυσκολία. Το πρόγραμμα λοιπόν προβλέπει ότι μετά από την δική μου σύντομη εισαγωγή μπορούν να πάρουν το λόγο είτε οι ευρωβουλευτές είτε οι βουλευτές των κοινοβουλίων. Πρέπει να δώσουμε μια κάποια τάξη στις ομιλίες αυτές. Νομίζω ότι έχει ίσως ήδη διανεμηθεί ένα χαρτί. Μπορείτε να γράψετε το όνομά σας και να ζητήσετε να μιλήσετε. Μπορείτε να το δώσετε στην γραμματεία που βρίσκονται εδώ αριστερά. και όταν συγκεντρώσουμε τον κατάλογο αυτών που θέλουν να πάρουν το λόγο θα δούμε τι χρόνο θα έχει ο καθένας στη διάθεσή του έτσι ώστε να εκφραστούν όλοι οι βουλευτές στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου χρόνου. Με ένα μέγιστο χρόνο δηλαδή παρέμβασης του καθενός. Νομίζω ότι θα κλείσουμε τη σημερινή, την πρωινή συνάντηση με ένα γεύμα εργασίας οι βουλευτές θα βρεθούν σε ένα γεύμα που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά τη διάρκεια του γεύματο αυτού μπορούμε με απόλυτη ελευθερία να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την συζήτηση γύρω από την ενιαία εκλογική διαδικασία η τροποποίηση της πράξης του 76, της 20 Σεπτεμβρίου του 76, η οποία είναι σήμερα ενισχύ και η πρόβλεψη μιας ενιαίας εκλογικής διαδικασίας προβλέπεται στο 2.23 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει την δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλει ένα σχέδιο, ένα προσχέδιο μάλλον. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο εμείς θα μπορούσαμε να μην κάνουμε. Εξ αρχής δηλαδή ήδη από το 1951 όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα η συνθήκη έδινε την δυνατότητα να υπάρξει ένας εκλογικός νόμος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τότε. Στη συνέχεια έγιναν πάρα πολλές απόπειρες με διαφορετικά αποτελέσματα η κάθε μία. Και καταλήξαμε στην πρώτη άμεση εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1979 για πρώτη φορά. Κάποιες τροποποιήσεις έχουν υπάρξει στην πράξη του 1976 μετά το 2000 μετά από την έκθεση του κυρίου Αναστασόπουλου, του Αντιπροέδρου Αναστασόπουλου, αλλά οι τροποποίησεις δεν ήταν θα έλεγα αποφασιστικές. Τώρα πλέον έχει οριστεί ο Άντριου Νταφ σαν εισηγητής της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής για να προχωρήσει σε μια νέα κωδικοποίηση της πράξης του 1976 σχετικά με την ενιαία εκλογική διαδικασία. Όλοι μπορούν να διαπιστώσουν ότι γύρω από τις ευρωεκλογές υπάρχει μια προϊούσα θα έλεγα απομάκρυνση του Ευρωπαίου πολίτη. Στην Ιταλία ας πούμε το ποσοστό αυτών που ψηφίζουν έχει μειωθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια. Απαιτείται λοιπόν να προσπαθήσουμε να καλύψουμε και σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης σωστά τις ευρωπαϊκές εκλογές και θα πρέπει παράλληλα, δεν ξέρω αν ισχύει για όλες τις χώρες, αλλά σε πολλές σαν την Ιταλία θα ισχύει, ε, βλέπει ο κόσμος τις ευρωεκλογές όχι σαν ευρωπαϊκές, αλλά σαν εθνικές. Στην ουσία δηλαδή είναι καθρέφτης των εθνικών πολιτικών αντιπαραθέσεων. Θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια της προσπάθειας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας στους Ευρωπαίους πολίτες μέσω του εκλογικού συστήματος. Το προσχέδιο του συναδέλφου Νταφ προβλέπει μια περαιτέρω τροποποίηση της πράξης του 1976, μια συμπληρωματική συνθήκη η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ τις επόμενες, από τις επόμενες εκλογές ε, το 2014. Δεν είναι κάτι τέτοιο εύκολο γιατί υπάρχει και το θέμα της επικύρωσης από πλευρά των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη φάση εμείς εργαζόμαστε εντατικά και νομίζω ότι και αυτή εδώ η συνάντηση θα βοηθήσει έτσι ώστε να εμβαθυνθεί η συζήτηση έχω μακρηγορήσει, ζητώ συγγνώμη και θα ήθελα να παρακαλέσω τον συνάδελφο Νταφ να πάρει το λόγο και να κάνει μια νέα εισαγωγή στην ε, συζήτησή μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σας λόγια και για την περιγραφή του πλαισίου της εκθέσεως με τόσο σαφή τρόπο. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η συνεργασία μεταξύ βουλευτών σαν φιλής είναι εξαιρετικά σημαντική αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσουμε την λαϊκή νομιμοποίηση της Ένωσης. Όπως ξέρετε, τα τελευταία 10-12 χρόνια διαμορφώνουμε αλλαγές συνθήκων που αύξησαν σαφώς την θεσμική νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εξαιρετικά δραματικό τρόπο. Ωστόσο, στην συνέλευση δεν σταθήκαμε σχεδόν καθόλου στα θέματα της λαϊκής νομιμοποίησης του Κοινοβουλίου. Και πιστεύω ότι ένα τμήμα της απογοήτευσης των πολιτών που επεδείχθηκε κατά τη διάρκεια των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων συνταγματικού χαρακτήρα προέκυψε από το γεγονός ακριβώς ότι δεν ασχοληθήκαμε με την σύνθεση και την εκλογική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξεκινώντας σήμερα την διαμόρφωση ισχυρότερων ε, δομών ε, διακυβέρνησης που επιβάλλουν υποχρεώσεις στους πολίτες ως φορολογούμενους και όχι μόνο ε, ως, ε, που επιβάλλουν εκλογικές ε, υποχρεώσεις πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στο να παραμένει το Κοινοβούλιο και λαϊκά δημοφιλές και να εκτιμάται από τους πολίτες. Το πακέτο των προτάσεων που υπέβαλα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει διανεμηθεί σε όλους σας. Δεν περιμένω να το διαβάσετε, να το έχετε διαβάσει όλο, διότι είναι πολύ μακρύ. Έχει μια μακρά ιστορική περιγραφή των εξελίξεων. της άμεση εκλογής του Κοινοβουλίου. Ωστόσο θεωρώ σημαντικό να καταλάβουμε το ιστορικό πλαίσιο Αυτόν που θέλουμε να πετύχουμε. Τέσσερα βασικά τμήματα περιλαμβάνει η πρόταση. Κατά σειρά προτεραιότητας θα προσπαθήσω να στη συνοψίσω. Πρώτον, υπάρχει το πρόβλημα των προνομίων και ασύλειών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή απολάβουμε, αν είναι σωστή αυτή η λέξη, ενός καθεστώτος που θεσπίστηκε το 1965 βάσει ενός πρωτοκόλου προνομίων και ασυλιών που υποχρεώνει τους Ευρωβουλευτές και το Κοινοβούλιο να υπάγονται στην αντίστοιχη εθνική τους νομοθεσία. Τούτο δημιούργησε μια σειρά προβλημάτων συνοχής και συνέπειας σε ό,τι αφορά το ισότιμο καθεστώς των ευρωβουλευτών ως τμήμα του πακέτου θέλουμε να αναθεωρήσουμε την, το πρωτόκολλο αυτό του 1965. Το δεύτερο ζήτημα αφορά το πρόβλημα των πολιτών της Ένωσης που κατοικούν σε άλλη χώρα και όχι την χώρα της ηθαγένειάς τους. Η Eurostat εκτιμά ότι γύρω στα 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες είναι μόνιμοι κάτοικοι σε άλλη χώρα πλην της δικής τους. Η συνθήκη όπως γνωρίζετε αναφέρει ότι οι πολίτες που κατοικούν σε κράτος άλλο αυτού της ηθαγένειάς τους πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στις εκλογές για την Δημοτική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην πράξη αυτό φαίνεται ότι αποτελεί, αποδεικνύεται μάλλον ότι είναι προβληματικό ως προς την υλοποίησή του. Δηλαδή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη η διάταξη αυτή της συνθήκης, καθότι υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά προσκόμματα σε πολίτες που θέλουν είτε να ψηφίσουν είτε να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όλο ένα και περισσότερο υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία πολιτικής ε, θέσης προς κομμάτων σε ορισμένα κράτη από ε, ορισμένες κρατικές αρχές που επιδιώκουν να παρεμποδίσουν το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να απολάβουν όλων των δικαιωμάτων που δικαιούνται. Όπως γνωρίζετε υπάρχει και μια οδηγία 93 κάθετος 109, η οποία προσπάθησε να υλοποιήσει αυτή την διάταξη της συνθήκης που είχε ξεκινήσει, που είχε πρωτοεισαχθεί με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Η Επιτροπή προσπάθησε να αναθεωρήσει την διαδικασία για να απλοποιήσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες που θα επιτρέπουν στους πολίτες Ένωσης να μπορούν να, τύχουν δημοκρατικής, ε, να έχουν τη δημοκρατική συμμετοχή που δικαιούνται. Αλλά η απόφαση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη στο Συμβούλιο και ως τμήμα ενός ευρύτερου πακέτου εκλογικών μεταρρυθμίσεων θα ήλπιζα ότι η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει εκ νέου το ζήτημα παρουσιάζοντας μια πιο ρηξικέλευτη πρόταση που θα αντικατοπτρίζει πιστότερα τις θεσμικές απαιτήσει στην εκλογική νομοθεσία. Το τρίτο από τα τέσσερα μεγάλα στοιχεία αφορά την κατανομή των ευρών μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ένωσης στο υφιστάμενο κοινοπούλιο. Όπως γνωρίζετε, το πρέπει να διανεμηθούν 751 έδρες μεταξύ 27 κρατών βάσει της αρχής της φθήνουσας αναλογικότητας που περιγράφει και αναφέρει συνθήκη. Υπάρχει πολιτική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου να οριστεί η έννοια της αρχής της φθήνουσας ε, αναλογικότητας. Συγγνώμη. Δεν περιέχεται ακόμα σε ένα νομοθετικό κείμενο. Αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο υπάρχουν εννέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η αρχή αυτή δεν τηρείται και δεν νομίζω ότι είναι σωστό το ίδιο το Κοινοβούλιο να παραβιάζει τη συνθήκη. Επίσης, είναι σημαντικό μετά την προσθήκη των 18 μελών του Κοινοβουλίου που θα γίνουν μέλη του Κοινοβουλίου μετά την θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Θα υπάρχουν ακόμα πέντε περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της συνθήκης. Κάτι απαράδεκτο κατά την άποψή μου. Επίσης πιστεύω ότι το σύστημα διανομής ευρών μεταξύ κρατών στο παρελθόν ήταν χαοτικό, αδιαφανές και απετέλεσε αιτία πολιτικών συγκρούσεων ασύλληπτων στο πάθος τους ε, και ήταν ένα μέρος των παζαριών μεταξύ κρατών με τελείως ε, αδιάφανο τρόπο στα πλαίσια ευρύτερων δια κυβερνητικών διαπραγματεύσεων που θυμίζει περισσότερο ε, ρουλέτα παρά συνταγματικές διαπραγματεύσεις. Μέχρι ότου βρεθεί μια μαθηματική φόρμουλα συγγνώμη, που θα ρυθμίζει την διανομή των θέσεων ε, των 751 ευρών, 51 κάθε πέντε χρόνια και που θα φέρει το επιχείρημα τη συζήτηση από την ε, πολιτικά διαπραγμάτευση στην πολιτική διαπραγμάτευση δεν θα ολοκληρωθεί, δεν θα λυθεί το ζήτημα. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να συμφωνήσουν και οι ίδιοι μαθηματικοί για την φόρμουλα που θα επιλεγεί και το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει ένα ρόλο σε ένα εγχείρημα στο οποίο καθηγητές εφαρμοσμένων μαθηματικών που είναι ειδικοί στο θέμα αυτό θα κληθούν να συμφωνήσουν με μία εξίσωση που θα είναι αποδεκτή και από μας. Το τέταρτο και προφανώς πιο σημαντικό και και η μεγαλύτερη αλλαγή που προτείνω είναι να δημιουργηθεί μία πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια για την εκλογή επιπλέον 25 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η, τα ψηφοδέλτια θα υποβάλλονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που υπάρχουν, αλλά παρότι δεν είναι πλήρως αναπτυγμένα πολιτικά κόμματα υπό την έννοια που το καταλαβαίνουμε στο ε, εθνικό πλαίσιο. Η απουσία ουσιαστικών πολιτικών κομμάτων από την ευρωπαϊκή πολιτική ζωή είναι ένα βασικό θεμελιώδες ελάττωμα Και η διαμόρφωση τέτοιων κομμάτων, ε, τέτοιων εκλογικών συνδυασμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα βοηθήσει να καλυφθεί αυτό το κενό. Κάθε ψηφοφόρος λοιπόν το 2013 θα παίρνει δύο ψηφοδέλτια μπαίνοντα ε, στο εκλογικό κέντρο. Το πρώτο για την εθνική ή περιφερειακή ε, εκλογική περιφέρειά του και ένα δεύτερο με το ψηφοδέλτιο των 25 υποψηφίων που επιλέγουν στη σειρά που θέλουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Το σύστημα που προτείνω είναι ένα ημιανοιχτό σύστημα με ψήφο προτίμηση ούτως ώστε ο ψηφοφόρος να μπορεί να επιλέξει είτε να ψηφίσει τη λίστα όπως την θέτει το πολιτικό κόμμα ή να επιλέξει να δώσει την προτίμησή του σε έναν συγκεκριμένο υποψήφιο. Θα σκεφτόμουν ότι ο διάδοχος του πρόεδρου Μπαρόζο στην Προεδρία της Επιτροπής θα πρέπει να συμπεριλαμβανόταν να συμπεριλαμβάνεται μάλλον σε αυτή την υπερεθνική λίστα. Έγινε μεγάλη, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση μεταξύ των ε, πολιτικών κομμάτων για την προσπάθεια να βρουν ε, ε, πρωταθλητές που θα προωθήσουν τις θέσεις τους στις προηγούμενες ευρωεκλογέ. Το να βρεις ωστόσο έτσι θεωρητικά έναν πρωταθλητή, ιδίω όταν ο πρωταθλητής αυτή, αυτός ήταν ένας πρώην, ένα πρώην ηγετικό, μια πρώην ηγετική προσωπικότητα σε ένα κράτος μέλος, πρώην είναι πρωθυπουργός ή τέλος μεγάλη πολιτική προσωπικότητα, θα συνεχίσει να είναι ε, απίθανο. Διότι οι μεγαλόσχημοι δεν θέλουν οι ίδιοι να σταθούν, να κατεβούν σε εκλογές και να κινδυνεύσουν να ιτηθούν. Εάν υποχρεώσουμε τους πρωταθλητές αυτές να επιδιώξουν μια θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το όλο εγχείρημα θα προσγειωθεί πολιτικά και θεσμικά στην παραδοσιακή κοινοβουλευτική κουλτούρα των εκλογών. Τρία από τα τέσσερα θέματα, το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες, ο μαθηματικός τύπος για την ε, κατανομή των βουλευτών και η διεθνική λίστα, το διεθνικό ψηφοδέλτιο θα απαιτήσουν αλλαγή της συνθήκης. Και οι συνάδελφοι ε, λένε ότι έχουν πάθει μία συνθηκοκόπωση. Λυπούμε γι' αυτό. Ε, κανείς δεν μου είπε ότι θα έπρεπε να είμαι κουρασμένος όταν ε, ήλθα στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ωστόσο όλοι ότι προφανώς ε, οι αλλαγέ συνθήκων αποτέλεσε κινητήρια δύναμη και της ενοποίησης και της ε, εμβάθυνσης της δημοκρατίας. Πιστεύω ότι εμείς που ασχολιόμαστε κυρίως με συνταγματικά θέματα πρέπει να υπενθυμίσουμε την ιστορική λειτουργία των ε, αλλαγών των συνθήκων για την πρόθεση της ενοποίησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξει. Όπως ξέρετε το Κοινοβούλιο πρέπει να ξεκινήσει ε, ε, ε, το ίδιο της διαδικασίας μεταρρύθμιση εφόσον η Επιτροπή δεν τολμά να κάτι τέτοιο. Εάν το, το Κοινοβούλιο σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες μέχρι το Δεκέμβριο και να παραπέμψει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου ο κύριος Βαν Ρόμπερ έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να επανεξετάσει το, το φάκελο αυτό. και να μείνει στα χέρια του και όχι στα χέρια της, ε, ε, ε, των αλλαγών του τρίο, των, ε, της προεδρίας του Τρίου Όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπή στο ξεκίνημα, ε, θα γίνει, πρέπει να γίνει μια συζήτηση εδώ που θα προκαταλάβει την διακυβερνητική διάσκεψη ή τη συνέλευση. Η δική μου προτίμηση είναι να υπάρξει μια συνέλευση. Προφανώς ε, τούτο προέρχεται από την παλιά εμπειρία μου ε, συμμετοχή στις δύο προηγούμενες συνελεύσεις που πρέπει να σας πω ότι μου άρεσαν πάρα πολύ και τις απόλαυσα. Στη συνέλευση αυτή, στην οποία θα μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ε, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Εθνικά Κοινοβούλια, εκπρόσωποι Πρωθυπουργών και που θα συζητήσει αυτό το πακέτο, θα αποτελέσει ένα γόνιμο και χρήσιμο εργαλείο. Με ευρύτερη νομιμοποίηση από την απλή παραπομπή του θέματος από το Κοινοβούλιο στη διακυβερνητική διάσκεψη, ωστόσο παραμένω ανοιχτός για κάθε πρόταση διαδικαστικού χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και το χρονικό πλαίσιο δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις. Αν θέλουμε η μεταρρύθμιση να ολοκληρωθεί έγκαιρα για να λειτουργήσει το 2014, θα πρέπει να πατήσουμε γκάζι. Ίσως ε, μίλησα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μην ήμουν ωστόσο ε, χωρίς ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σαφήνεια με την οποία μιλήσατε και την περιεκτικότητα της ομιλής σας. Ε, διευκρινίσατε σε τρία θέματα, ένα περίπλοκο θέμα. Υπάρχουν και βεβαίως άλλα δευτερεύοντα ε, τα οποία υπάρχουν στο εγγραφό σας και αναφερθήκατε και εσείς σε αυτά. Νομίζω όμως ότι σήμερα η παρέμβαση σας αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα να διευκρινίσετε τα τέσσερα θέματα από τον οποίο θα ακολουθήσει η συζήτηση. Μέχρι τώρα έξι άτομα έχουν ζητήσει να παρέμβουν και βεβαίως ε, όποιος επιθυμεί να παρέμβει μπορεί ακόμα ε, να, το, να ζητήσει το λόγο. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουν ζητήσει τέσσερις εθνικοί βουλευτές και δύο ευρωβουλευτές να παρέμβουν. Και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο πρώτα σε δύο εθνικούς βουλευτές, έναν ευρωβουλευτή, μετά θα ακολουθήσουν πάλι δύο εθνικοί βουλευτές και ο δεύτερος ευρωβουλευτής. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, αν κάποιος ε, θέλει να παρέμβει, ε, ακόμα μπορεί να ζητήσει το λόγο. Θα θα λοιπόν να δώσω το λόγο ε, στον συνάδελφο από την Φινλανδία, τον κύριο Γιωάννης Κόσκινεν. Πρόεδρε, Αυτό το έγγραφο εργασίας ε, του κυρίου Νταφ, το σχέδιο της ε, έκθεσης, είναι πραγματικά ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Υπάρχει ε, στο έγγραφο αυτό μια ολόκληρη σειρά πραγμάτων που και εμείς μπορούμε να στηρίξουμε ως Φινλανδία. Βεβαίως πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά το θέμα αυτό και κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει τις προτάσεις μας να τις συμπεριλάβουμε ε, σε έναν κατάλογο που να αφορά όλους τους ε, Ευρωπαίους. Γιατί με τον τρόπο αυτό ε, θα αλλάξει και η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, όσον αφορά στο εκλογικό δίκαιο, στους ε, δημοκρατικούς κανόνες ε, για τις εκλογές και για τις ε, προϋποθέσεις. Βεβαίως όλα αυτά τα υποστηρίζω. Θα ήθελα όμως να το σκεφτούμε λιγάκι το θέμα. Και κατά τα άλλα νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε το κατά πόσον ε, θα πρέπει ή χρειαζόμαστε υπερεθνικά δικαιώματα και ασυλίες. Όσον αφορά, ε, παραδείγματο χάρη, στην ε, προστασία του περιβάλλοντος, εκεί μπορούμε να σκεφτούμε το κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο όπως και τα εθνικά κοινοβούλια. Δηλαδή να εκπονηθούν κανόνες για καλές ε, ευρωπαϊκές πρακτικές σχετικά με το θέμα αυτό πάντα. Όσον αφορά τη χρονική στιγμή εκλογών, ο Μάιος θεωρώ ότι είναι κατάλληλη ημερομηνία, διότι Μάιος ε, δεν είναι ακόμα περίοδος εκλογών. Ε, μέχρι τώρα, τον Ιούνιο, όταν λάμβαν χώρα εκλογές, τουλάχιστον στις σκανδιναβικές χώρες, είχαμε διακοπές. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά πραγμάτων που θέλω να σκεφτώ περαιτέρω. Και όσον αφορά το θέμα του επιπρόσθετου αριθμού βουλευτών, θα ήθελα παρακαλώ να μου επιτρέψετε να το σκεφτώ λιγάκι αυτό. Βεβαίως όλο αυτό το θέμα δεν πρέπει να ερμηνευθεί αρνητικά. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ε, ευχαριστούμε καταρχήν τον κύριο Κόσκινεν ε, και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Λόρδο Μπόουνες από το ε, Κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που καλέσατε τα μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ντάφ για την ε, έκθεσή του. Όπως ε, και ο συνάδελφός μου από τη Φιλανδία είπε και για μας και το ίδιο. Εμείς δεν έχουμε τοποθετηθεί επ' αυτών των προτάσεων. Αλλά κατανοώ βέβαια την επιθυμία του κυρίου Νταφ, την οποία συμμεριζόμαστε όλοι μας. Επιθυμούμε δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη ε, συμμετοχή ε, των πολιτών στις ευρωπαϊκές εκλογές, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα έχει μεγαλύτερη σημασία για όλου μα. Εσύ ο ίδιο, ε, κύριε Πρόεδρε, Υπενηχθήκατε ένα πρόβλημα, το ότι οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζονται ως ευκαιρία για να εκφραστεί η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια με την οποιαδήποτε εθνική κυβέρνηση και κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας για το Ευρωκοινοβούλιο λίγα θέματα συζητώνται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε σε βάθος. Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια και οι εθνικές κυβερνήσεις ε, δεν επιθυμούν να συζητήσουν ε, τον αυξανόμενο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τούτο λοιπόν σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία στα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, στο μυαλό των ανθρώπων να ε, εμπεδοθεί αυτός ο διακριτός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπορώ βέβαια να ομιλήσω εξ ονόματος των υπολείπων 26 κρατών, όμως ε, αναμφίβολα τέτοιου είδους ε, ηγετικός ε, ρόλος δεν υπήρξε στο, Ευρωπαϊκό, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατανοώ βέβαια ε, το τι επικρατεί στα κράτη-μέλη, όμως εκεί προβλέπω προβλήματα γιατί κάθε κράτος μέλος για τους δικούς του λόγους έχει τη δική του εκλογική παράδοση. Ε, δίνει ιδιαίτερη σημασία στις εκλογικές περιφέρειες, στην ημερομηνία εκλογών και δεν νομίζω βέβαια αν υπάρξει μια πανευρωπαϊκή μερινομηνία ότι αυτό θα είναι αμφισβητήσιμο. Το 2014, κύριε Πρόεδρε, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος. Γνωρίζω ότι ο κύριος ε, Νταφ δεν υποφέρει από συμβασοκόπωση, αλλά ε, αυτό όμως ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το ισχυστούμε και για τα εθνικά κοινοβούλια. Εγώ συμμερίζομαι ε, το δυναμισμό του όσον αφορά στα προβλήματα που υπάρχουν. Αν λοιπόν θέλουμε να προχωρήσουμε, πραγματικά θα πρέπει να έχουμε ε, μια πιο ρεαλιστική ε, προσέγγιση, έστω και λιγότερο φιλόδοξη, ως προς το χρονοδιάγραμμα. Να αναζητήσουμε την υποστήριξη των κρατών μελών, των μελών εθνικών κοινοβουλίων και ας μην ξεχνάμε και των εθνικών πολιτικών κομμάτων. Η εκστρατεία για τέτοιου είδους αλλαγές αναπόφευκτα θα λάβει χώρα, κατά τη γνώμη τουλάχιστον, στα κράτη-μέλη. Και ε, οι εθνικές κυβερνήσεις, τα εθνικά κοινοβούλια και τα εθνικά πολιτικά κόμματα ε, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. για να εξηγήσουν αυτές τις ε, αλλαγές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί είναι υπερβολικά, υπερβολικά αισιόδοξοι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν συμμερίζουμε πολλές από τις φιλόδοξες απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Νταφ. Ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρθηκαν κάποιες ε, δυσκολίες, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο ε, παραμένουμε αδρανείς. Άρα δηλαδή το πιο σημαντικό από όλα είναι να αντιμετωπίζει κανείς τις προκλήσεις. Ο συνάδελφος κ. Σόπφλινγκ, ευρωβουλευτής, έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Ντάφ ε, ως ε, προς τις φιλόδοξες απόψεις του. Αλλά επιτρέψτε μου καταρχήν να πω ότι εγώ μιλάω ως ε, σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ για την έκθεσή του. Ε, συμφωνώ και επαυξάνω ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτω από αυτό το πρίσμα βέβαια η συνεργασία όπως αυτή που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στα εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι, ε, είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Και ελπίζω σήμερα από τη συζήτησή μας να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται σε μία σειρά θεμάτων που έχουν σχέση με τις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών. Όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης του κυρίου Νταφ, εδώ συμφωνώ απόλυτα, ε, πράγματι εξετάζουμε το θέμα της ε, υπηκότητας, ε, την υπηκότητα, την θαγένεια μάλλον, πώς μπορούμε να την ε, αντιμετωπίσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ε, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο. Εγώ γνωρίζω ότι η διπλή ηθαγένεια δεν αναγνωρίζεται. Έτσι λοιπόν αυτά που λέει ο κύριος Νταφ ε, είναι ιδιαίτερα θετικά. Το θέμα είναι η ταχύτητα. Θα ευχόμουν να μην ήταν έτσι. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα όσο θα επιθυμούσε ο κύριος Νταφ. Και πάνω απ' όλα, νομίζω εκφράζω σε μεγάλο βαθμό ε, τις απόψεις του πολιτικού μου κόμματος, αλλαγή συνθήκης. Σε αυτή τη φάση ε, είναι εξωπραγματικό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Ευρώπη, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνιολογικά. Νομίζω λοιπόν ότι το περιεχόμενο της έκθεσης του κυρίου Νταφ βεβαίως και είναι ευκταίο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με τον υπερεθνικό κατάλογο, αλλά η χρονική στιγμή δεν βολεύει. Εκεί διαφωνούμε και εκεί θα εκφράσουμε κάθετα τη διαφωνία μας. Μου αρέσει βέβαια η ιδέα της ε, συνέλευσης, ε, του να συνέρχονται οι άμεσα εμπλεκόμενοι, αλλά επαναλαμβάνω όχι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ενδέχεται λοιπόν η λύση να είναι πράγματι να έχουμε μία μακρά ε, προεκλογική εκστρατεία σε βάθος συζητήσεις εδώ και αλλού για αυτό το γενικότερο πρόβλημα το σκεπτικό αν θέλετε του να παρισφρήσει η ευρωπαϊκή διάσταση στη συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα, απέχει, δεν υπάρχει αυτή η διάσταση αυτή τη στιγμή, όμως με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, το Κοινοβούλιο έχει μεγάλη νομοθετική εξουσία και θεωρώ ότι απλά δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το γεγονός ότι ε, μειώνεται η προσέλευση στις εκλογές, αυτό είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι οι πολίτες δεν ταυτίζονται με αυτά που διαδραματίζονται στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το θέμα ε, τα επιχείρηματα του κυρίου Νταφ είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω πολλοί εθνικοί βουλευτές όταν θα επιστρέψουν στις ε, πατρίδες τους ε, θα παρουσιάσουν πολλά από αυτά που είπαμε, όχι απαραίτητα δικά μου, αλλά έστω όλα τα υπόλοιπα που θα λεχθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Μπεν Φαγιό, ο οποίος είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι κάθε φορά επιστρέφω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ιδιαίτερα στις εργασίες της ε, συνταγματικής αυτής επιτροπής. Η Επιτροπή σας είναι πάντα πρωτοπορία στην επεξεργασία θέσεων για τα θεσμικά όργανα και τις συνθήκες. Η φάση την οποία βιώνουμε εκπλήσει ορισμένου Λίγο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ξεκινάμε πάλι συζητήσεις θεσμικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος. Εγώ είμαι υπέρ, είμαι ο παδός φανατικός της κοινοβουλευτικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι η ενίσχυση αυτής της διάστασης θα οδηγήσει σε περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη. Όταν βλέπει κανείς τα ποσοστά συμμετοχής στις ευρωεκλογές, διαπιστώνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για την δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως εκ τούτου κάτι θα πρέπει να γίνει. Είμαι υπέρ της ιδέας να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα συνέλευση θα έλεγα, έτσι όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαφώνας, όχι τόσο για να συζητήσουμε κάποια θέματα τα οποία αφορούν αλλαγές στην ίδια τη συνθήκη, αλλά για να μπορέσουμε να ορίσουμε σωστά το θέμα του δημοκρατικού ελλείμματος. Μου δημιουργείται η αίσθηση ότι όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν μια σύγχυση για το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις αυτές και πρέπει με κάποιο τρόπο το ε, έλλειμμα το δημοκρατικό να το καλύψουμε. Ο Άντζιου Ντάφο συνήθως μας έδωσε ένα εξαιρετικό κείμενο. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Θα ήθελα να πω ότι ακόμα και η μετάφραση είναι εξαιρετική. Η εισαγωγή επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει ακριβώς την πορεία που ακολούθησε η δημοκρατία στην Ευρώπη μία πορεία προς ένα ισχυρό και πολιτικά σημαντικό βαρύνων κοινοβούλιο. Γύρω από τις προτεραιότητες τις οποίες σημειώνει ο Αντζουνταφ, καταρχάς σχετικά με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών που δεν είναι από την χώρα στην οποία κατοικούν. Εγώ προέρχομαι από μία χώρα, το Λουξεμβούργο, όπου το 40% των πολιτών που παραμένουν εκεί είναι ε, εκτός, ε, είναι, δεν έχουν καταγωγή, δεν είναι πολίτες του Λουξεμβούργου. Είναι μια χώρα το Λουξεμβούργο για τον οποία υπήρξε εξαίρεση όπως θυμάστε στη συνθήκη του Μάστριχτ για τις χώρες δηλαδή στις οποίες άνω του 20% των πολιτών δεν είναι πολίτες της χώρας αυτής μπορούν οι χώρες αυτές λοιπόν να πετήσουν σαν παράδειγμα πριν από τη δυνατότητα πρόσβασης στο δικαίωμα ψήφου μία χρονική περίοδο παραμονής. Μετά από 15 χρόνια εμπειρίας από τη λειτουργία αυτής της εξαίρεσης, νομίζω ότι δεν ήταν απαραίτητη, τουλάχιστον δεν είναι πλέον απαραίτητη. Η πλειοψηφία της πολιτικής τάξης της χώρας μου δεν το πιστεύει αυτό. Εγώ προσωπικά όμως θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το απαραίτητο η εξαίρεση αυτή. Διαπιστώσαμε κάτι το ενδιαφέρον στις τοπικές εκλογές, στις δημοτικές εκλογές. Οι μη Λουξεμβούργοι πολίτες που παραμένουν στην χώρα αυτή, είτε από τρίτες χώρες είτε από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκεί συμμετέχουν όλο και περισσότερο στις τοπικές δημοτικές εκλογές. Βέβαια αυτό γίνεται εξελικτικά, σταδιακά, σε διαφορετικές φάσεις. Αντίθετα στις ευρωεκλογέ το πράγμα λειτουργεί διαφορετικά. Στις ευρωεκλογέ διαπιστώνει κανείς ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν είναι Λουξεμβούργοι αλλά ζουν στο Λουξεμβούργο έχουν την τάση, λέω τάση έτσι δεν είναι άσπρο ή μαύρο, έχουν την τάση να πηγαίνουν να ψηφίζουν ή να ψηφίζουν γενικότερα στην δική τους χώρα προέλευσης και όχι τόσο στην χώρα όπου ζουν, δηλαδή στο Λουξεμβούργο. Πρέπει να το σημειώσετε αυτό. Αυτό δείχνει ότι πράγματι στα πλαίσια της πολιτικής δραστηριότητας των Ευρωπαίων πολιτών υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκλογική του συμπεριφορά. Ακόμα και αν ζουν οι άνθρωποι αυτοί επαναλαμβάνω σε άλλη χώρα από τη χώρα προέλευσή τους. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσουμε όταν συζητάμε για την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Στο κείμενο του Άντζιου Νταφ είδα ότι ζητά να υπάρξει μια νέα διαδικασία ή θα μπορούσε να ζητήσει μια τέτοια νέα διαδικασία λέγοντας ότι θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα ψήφου όχι μόνο σε τοπικές και ευρωπαϊκές αλλά και στις εθνικές βολευτικές εκλογές στους Ευρωπαίους πολίτες που δεν κατάγονται από τη χώρα στην οποία παραμένουν. Όπως γνωρίζω πάντως τη χώρα ε, ε, τη δική μου κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό. Το πρόβλημα είναι πολιτικό, είναι ένα πρόβλημα μιας κοινωνίας στην οποία το 40% δεν αποτελείται από λουξεμβούργιους. Πρόκειται για ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο συζητιέται ε, επανειλημμένα, έχει συζητηθεί επανειλημμένα και ε, καλό θα ήταν να ακούσουμε και τις απόψεις των υπολείπων βουλευτών. Μία άλλη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω γύρω από αυτήν την, αυτόν τον εκλογικό, το, το, το ψηφοδέλτιο, το διεθνικό ουσιαστικά, το οποίο προτείνεται. Δεν είναι πρώτη φορά που προτείνεται κάτι τέτοιο. Ήδη από τη δεκαετία του 90 είχαν υπάρξει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έκαναν αυτή την πρόταση. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ της ευρωπαϊκής διάστασης των πολιτικών κομμάτων, του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος. Όταν ήμουν ευρωβουλευτής, στα πλαίσια της προετοιμασίας της συνθήκης της Λισαβόνας, της του Μάστριχτ συγγνώμη, είπα ότι δεν είναι σωστό να υπάρχουν κοινοβουλευτικέ ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά να μην υπάρχει πολιτικό κόμμα στο οποίο να αναφέρεται η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Συνεπώς και στα πλαίσια της συνθήκης της, ε, του Μάστριχτ ορίσαμε για την δυνατότητα δημιουργίας των ευρωπαϊκών κομμάτων. Η εξέλιξή τους όμως με έχει απογοητεύσει. Τα κόμματα αυτά στην ουσία είναι κομματικοί οργανισμοί μεν των κομμάτων που τα συναποτελούν. Δεν είναι πραγματικά πολιτικά κόμματα. Είμαι λοιπόν πολύ διστακτικός γύρω από τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα. Προσωπικά δεν νομίζω ότι θα προσφέρει ε, η συνέχιση αυτής της προσπάθειας ε, κάτι το ιδιαίτερο στα πλαίσια της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Μπορεί να δημιουργήσει αν θέλετε ένα κάποιο σοου τηλεοπτικό λόγω της παρουσίας πολιτικών προσωπικότητων. Από την άλλη όμως δεν θα παράγει ενδιαφέροντες ευρωβουλευτές. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να υπάρχουν ευρωβουλευτές εργατικοί που να αντιπροσωπεύουν και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εκλογέων τους. Εγώ εδώ θα έβλεπα μάλλον περισσότερο μια θα έλεγα απόπειρα πιθανότητα δημιουργίας διασυνοριακών εκλογικών περιοχών. Εμείς στο Λουξεμβούργο συνεργαζόμεθα και οικονομικά και πολιτικά με τις όμορες περιφέρειες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Βελγίου. Και εκεί η Ευρώπη αποτελεί μια πραγματικότητα η οποία βιώνεται καθημερινά. Ο κόσμος μετακινείται σαν να μην υπήρχαν σύνορα. Ως εκ τούτου εκεί η εκλογική περιφέρεια η ευρωπαϊκή βρίσκει την δικαιολογία της αν θέλετε. Και όχι ε, κάτι το θεωρητικά μεγάλο που θα καλύπτει 27 χώρες κτλ. Δεν έχω άλλα να πω σε αυτή τη φάση. Μπορώ να κάνω και άλλα σχόλια βέβαια για το κείμενο του Νταφ Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει η συζήτηση για το δημοκρατικό έλλειμμα, για την πιθανότητα βελτίωσης του δημοκρατικού διαλόγου στα πλαίσια μιας νέας ας πούμε συνάντησης, συνέλευσης. συνέλευσης. Ευχαριστώ τον κύριο Μπενφαγιό. Ο κύριος Φαρούτζια, Άντζελο Φαρούτζια από τη Μάλτα, ορμόμενος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Νταφ για την έκθεσή του και νομίζω ότι τα σχόλιά του έρχονται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Όπως είπε και ο πρόεδρος, προέρχομαι από τη Μάλτα και η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας θα πρέπει να τηρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών και άλλες αρχές για να μπορέσει η συνθήκη να υλοποιηθεί. Μιλούμε εδώ για το πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ε, ευρωπαϊκή δημοκρατία. Όταν μιλάμε για δημοκρατία θα πρέπει να δούμε ότι τα δικαιώματα των ε, ψηφοφόρων, των ατόμων που έχουν το δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Σε μια χώρα μικρή, όπως η χώρα μου, η Μάλτα, όπου οι εκλογές κερδίζονται από μερικές εκατοντάδες ψήφων και μάλιστα στις τελευταίες ε, εκλογές το 2008 και στις προηγούμενες ευρωεκλογές η, απόσταση μεταξύ των, η απόκληση μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων ήταν λίγες εκατοντάδες ψήφων. Αυτό είναι διαφορετικό προφανώς από το τι συμβαίνει στα μεγάλα κράτη-μέλη. Γιατί σα τα λέω αυτά τώρα. Γιατί αν υπάρξει, αν δεν αλλάξει σοβαρά το εκλογικό σύστημα και στη Μάλτα για παράδειγμα είμαστε πίσω στην εκλογική μεταχείριση, ε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που παρουσίασε ο κύριο Νταφ. Πρέπει να υπάρξει μεγάλη εκλογική μεταρρύθμιση πριν προχωρήσουμε στην μεταρρύθμιση του κύριου Νταφ. Για παράδειγμα, στη Μάλτα και κάθε χώρα έχει τη δική της εκλογική νομοθεσία. Ε, στη Μάλτα κάθε, άτος, κάθε άτομο για να ψηφίσει πρέπει να έχει ε, ταυτότητα. Πρέπει να παρουσιάσει την ταυτότητά του για να ψηφίσει. Έτσι γίνεται ο έλεγχος σε όλες τις εκλογές στη χώρα μου. Ε, δημοτικές, εθνικές κλπ. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι έχει την ευθύνη του ότι το ίμιση των ταυτοτήτων έχει εκπνεύσει. Άρα περίπου οι μισοί ψηφοφόροι στη Μάλτα τυπικά δεν μπορούν να ψηφίσουν. Η έλεγχη λοιπόν της ταυτότητας των, των είναι δύσκολη. Επαναλαμβάνω, στη Μάλτα ο κόσμος, τα κόμματα αγωνίζονται πολύ για τις, σε κάθε εκλογή, ακόμα και για τις ευρωεκλογέ. Στη Μάλτα το ποσοστό της συμμετοχής στις εκλογές δεν είναι 30-40% αλλά 80 και 90% κατά συνέπεια. Πρέπει να εξετάζουμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση που μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε μικρές χώρες η μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος μπορεί να αλλάξει ριζικά την κατάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ενιαία, το ενιαίο εκλογικό ψηφοδέλτιο. Θα πρέπει το ενιαίο αυτό ψηφοδέλτιο να περιλαμβάνει μια ισορροπία εθνική και γεωγραφική. η αύξηση των μελών του Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των, δικό, των βουλευτών των εθνικών και ε, συμφωνώ σε αυτό με τον Φιλανδό συνάδελφο. Η παρέμβαση του συναδέλφου από τη Βουλή των Λόδων πρέπει να ε, είναι σωστή. Πρέπει να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και τις ε, απαιτήσεις που έχει κάθε κράτος μέλος και κάθε εθνική νομοθεσία. Αλλιώς δεν θα πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαρούτζα. Πάρα πολλοί άλλοι ζήτησαν το λόγο. Προτείνω να μην πηγαίνουμε πλέον με το ρυθμό δύο εθνικοί βουλευτές, ένας ευρωπαϊκός. Έτσι με, μια με ένα γρήγορο υπολογισμό θα πάμε ένας από εδώ, ένας από εκεί προσπαθώντας να υπάρχει μια αντιπροσώπευση και όλων των πολιτικών τάσεων για να μην αγνοήσουμε ακριβώς ε, καμία πολιτική ευαισθησία. Η κυρία Μπελία έχει το λόγο. Πρώτα ευχαριστώ. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφ, εισηγητή, για την ποιότητα της έκθεσής της, εξαιρετική ποιότητα, και να τον ε, διαβεβαιώσω για την υποστήριξή μας, την υποστήριξη των Ευρωπαίων οικολόγων στην πορεία που έχει ξεκινήσει και που σίγουρα θα προχωρήσει την ευρωπαϊκή δημοκρατία αφενός, θα φέρει δε κοντά τους πολίτες με το ευρωπαϊκό εγχείρημα αφετέρου. Να διευκρινίσω καταρχήν ότι έχουμε επίγνωση του ότι η λαϊκή νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι αρκετή. Δεν θα είναι αρκετή ε, για να εξασφαλιστεί μέσω της εκλογικής μεταρρύθμισης, αλλά θα συμβάλλει. Το ίδιο θα συμβάλλει και η πρωτοβουλία των πολιτών, αντικείμενο των απογευματινών συζητήσεών μας. Μπορεί να βελτιώσει την έννοια της ε, ευρωπαϊκής ηθαγένειας, αλλά δεν θα την αλλάξει ριζίκα. Αν θέλουμε, θεωρούμε ότι η πολιτική βούληση είναι να μειώσουμε την απομάκρυνση των πολιτών από την Ευρώπη, στη φάση αυτή θα έλεγα ότι κανένα εργαλείο ή καμία παρέμβαση δεν πρέπει να αγνοηθεί. Πιστεύω ότι η έκθεση DAF, η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής εκλογικής διαδικασίας μπορεί κάλλιστα να συμβάλλει σε αυτό. Θα ήθελα να σας υποβάλω παρατηρήσεις και σκέψεις σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, οι ευρωβουλευτές που θα εκλέγονται στην ενιαία ευρωπαϊκή λίστα. Συμμερίζομαι εν γέννη την θέση. Γιατί όμως 25? Γιατί μόνο 25 και όχι παραπάνω. Άλλη ερώτηση. Γιατί 25 πρόσθετοι βουλευτές. Για γιατί να μην υπάρξει ένας κανόνας που θα λέει μια ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στον αριθμό των υφιστάμενων βουλευτών. Ένα άλλο θέμα που μου προξένησε την προσοχή μου στην έκθεση. Αυτή η εκλογική αρχή όντως είναι αναγκαία αλλά κάτι που θα πρέπει να διευκρινίσουμε αφορά την ανάγκη να αποκτήσει αυτή η εκλογική αρχή πρώτον ανεξαρτησία και δεύτερον εχέγγυα πραγματικών δυνατοτήτων αμεροληψίας και ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων. Αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα επίλυσης εκλογικών διαφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη δυνατότητα βεβαίως να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τρίτο σημείο. Η ηλικία συμμετοχής στις ε, εκλογές. Η ηλικία των 16 για την μεν πρωτοβουλία πολιτών θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένη η ηλικία, αιτιολογεί την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ωστόσο, στην εκλογική διαδικασία μου δημιουργεί ερωτηματικά, διότι σημαίνει ότι δίνουμε πολιτικά και αστικά δικαιώματα σε πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα δικαιώματα αυτά δεν τα διαθέτουν στις περισσότερες περιπτώσεις στο εθνικό πλαίσιο. Για να τελειώσω. Είμαι πεπισμένη ότι μια εναρμόνιση των εθνικών ε, ε, εκλογικών συστημάτων είναι αναγκαία. Αναλογική εκπροσώπηση, μία μέρα για την εκλογή, συγκεκριμένη μέρα, θα είναι μέτρα που θα συμβάλλουν και στο να προχωρήσουμε την νομιμοποίηση του Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο Ισπανός γερουσιαστής Πέδρο Ραμόν Ντεμόρα έχει το λόγο τώρα. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Adesso, va, va bene. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εντάχει. Θέλω να συγχαρώ βεβαίω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον κύριο Ντάφ προσωπικά για την πρωτοβουλία του και για το γεγονό ότι κάλεσαν, καλέσατε του ε, εθνικού βουλευτέ. Θεωρώ και εγώ σημαντικό να υπάρχει συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων τη ε, Ένωσης ως εθνικός βουλευτής γερουσιαστή συγκεκριμένη περίπτωση. Λίγες μέρες μόνο γνωρίζω την πρωτοβουλία αυτή. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο δουλεύει το θέμα αυτό επί μακρόν. Είναι λογικό κατά συνέπεια να μην μπορώ να σας προσφέρω μια οριστική άποψη ούτε να εκφραστώ εξ ονόματος είτε του Κοινοβουλίου μου είτε των, α, της πολιτικής μου ομάδας στην Ισπανία. Υπάρχουν απόψεις αλλά δεν έχουμε ενιαία θέση. Με τη... Θα ήθελα ωστόσο να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να σας πω αυτά που λέω, διότι πιστεύω ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία που συγκατεύθυνση αυτή είναι ενδιαφέρουσα. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της νομιμοποίησης του Κοινοβουλίου με την ενίσχυση της δημοκρατικής διάστασης της Ευρώπης και μειώνοντας τις αποκλήσεις μεταξύ των εκλογικών διαδικασιών μεταξύ κρατών μελών είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που δεχόμαστε με θετικό τρόπο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα βεβαίως. Προφανώς είναι θεμελιώδους χαρακτήρα ο συντονισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταξύ το, του ευρωπαϊκού και των εθνικών εκλογικών συστημάτων. Διότι σκέφτομαι για παράδειγμα τις δυσκολίε που θα μπορούσε να οδηγήσει το γεγονός για παράδειγμα η εγγεγραμμένη το δικαίωμα ψήφου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι 16 από, για τους πολίτες από 16 ετών, ενώ για τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια να είναι από 18. Αυτό μπορεί να, υπά, να δημιουργήσει πρόβλημα. Ένας 16χρονος θα πει γιατί να ψηφίζω για εδώ και να μην ψηφίζω για εκεί. Είναι λοιπόν ζητήματα που σίγουρα θα απαιτούν μεγαλύτερη συμμετοχή, μεγαλύτερη, μεγαλύτερο συντονισμό, συγγνώμη. Η ιδέα ενός ε, πανευρωπαϊκού ψηφοδελτίου είναι εξαιρετική ιδέα ενισχύει την ιδέα της Ευρώπης. Έχω κάποιες επιφυλάξεις και δεν είμαι μόνος σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εκλογικές περιφέρειες στα κράτη-μέλη που έχουν πάνω από 20 εκατομμύρια κατοίκων. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα δημιουργούσε προβλήματα. Μπορού, θα μπορούσαν να ερμηνευθούν, να, να υπάρξουν και ερμηνείες ε, που δεν θα θέλαμε να υπάρχουν. Συμβαίνει, ξέρετε, πολλές φορές στην πολιτική να προσπαθούμε κάποιες φορές να κάνουμε δύο πράγματα που μπορεί να προκύψουν αντιφατικά εν τέλει. Είναι θετικό να μιλάμε για περισσότερη Ευρώπη. Αν μιλάμε όμως για περισσότερη Ευρώπη και ταυτόχρονα μιλάμε για περισσότερο περιφέρειες, ενισχύουμε το, το, συνολικό αλλά και το πιο περιορισμένο και αυτό μπορεί ενδεχομένω να δημιουργήσει αντιφάσει και προβλήματα. Πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά για να μην υπάρχουν και προβλήματα μεθοδιακού χαρακτήρα. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Πιστεύω ότι η ιδέα να υπάρξει μια συνέλευση είναι θετική γιατί θα μπορέσει να συζητήσει το θέμα αυτό και το Εθνικό Κοινοβούλιο. Κάποια πράγματα η αιτιολογική σκέψη J που αναφέρει, J δηλαδή, που αναφέρει ότι ε, πολίτες ε, που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος και μπορούν να ψηφίσουν ε, στις ευρωεκλογές είναι περιορισμένος. Αυτό δεν ισχύει παντού. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί πολίτες της, άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές και στις τοπικές εκλογές. Και έχουμε πολλούς δημοτικούς συμβούλους αλλοδαπούς. Στην περιοχή μου, τη Βαλένθια, έχουμε πολλούς, πολλά χωριά που έχουν περισσότερους κατοίκους μη Ισπανούς παρά Ισπανούς. Φαντάζομαι ότι και ο, συνάλλο... ο συνάδελφος ε, δίπλα μου είναι από τα Κανάρια νησιά. Μπορεί και εκεί να συμβαίνουν τα ίδια. Τι θέλω να πω. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια παντού στην Ευρώπη. Μπορεί στην ε, Βρετανία να υπάρχουν λίγοι Ισπανοί. Στην Ισπανία, ωστόσο, υπάρχουν πολλοί Βρετανοί πολίτε που μένουν εκεί και ασκούν το εκλογικό του δικαίωμα. Θα μπορούσαν να βγουν και δήμαρχοι σε κάποια χωριά που είναι πολύ οι αλλοδαποί. Αυτές είναι κάποιε πρώτε σκέψει μου, Πρόεδρε. Ευχαριστώ εκ νέου για την πρωτοβουλία σα και Πιστεύω ότι και στο μέλλον θα συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε όσο περισσότερο γίνεται τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για τον τρόπο με τον οποίο, χαίρομαι για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο τον συντονιστή των σοσιαλιστών στην ε, κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μιλώ ως συντονιστής της σοσιαλιστικής ομάδας στην ε, συνταγματική επιτροπή και εγώ με τη σειρά μου θέλω να καλωσορίσω θερμά τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ξεκινώ λέγοντας ότι συμμεριζόμαστε με τον εισηγητή κύριο Νταφ την αναγκαιότητα να ξεκινήσει αυτή η, αυτός ο προβληματισμός που περιλαμβάνει το κείμενο που συζητούμε. Πιστεύουμε ότι οι στόχοι που επιδιώκει για την τελειοποίηση του συστήματος ε, εκλογικής συμμετοχής και για την οικοδόμηση μιας καλύτερης ε, συσχέτισης πολιτών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένας ε, αναγκαίος στόχος δεδομένων των δεδομένων που εξηγήθηκαν εδώ και που δημιουργούν ανησυχίες για την σχέση αυτή πολιτών ένωσης. Θεωρούμε πολύ χρήσιμη τη συζήτηση που έχουμε μαζί σας και θεωρούμε πολύ αναγκαίο να σας ακούσουμε. Διότι, κατά πάσα πιθανότητα, η συζήτηση αυτή δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί χωρίς να ξέρουμε ε, σε βάθος τις πολιτικές θέσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και βεβαίως και των διαφόρων κομμάτων σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Θέλω να υπογραμμίσω κάποιες σκέψεις που έχουμε για τη συζήτηση αυτή ως πολιτική ομάδα και να, και μοιραστώ μαζί σας κάποιες αμφιβολίες. Πρώτον, θα ήθελα να φέρω ότι την αναφέρω ότι συμπίπτουμε σε πολλά σημεία με την έκθεση DAF. Δεν θα τι αναφέρω αυτέ. Έχουμε ωστόσο τέσσερις ομάδες σκέψεων που θέλουμε να μεταβιβάσουμε σε εσά. Πρώτον, οι εκλογικέ μεταρρυθμίσει που απαιτούν, μάλλον η μεταρρύθμιση που προτείνουμε, που απαιτεί εθνικές μεταρρυθμίσει των εκλογικών συστημάτων, είναι πάρα πολύ περίπλοκε. Για παράδειγμα, η αλλαγή τη ηλικία. Ε, σε κάθε χώρα, για τις ηλικίες δικαιώματος ψήφου σε κάθε χώρα. Η μεταρρύθμιση των εκλογικών περιφερειών σε κάθε χώρα. Η μεταρρύθμιση του εσωτερικού συστήματος κατανομής των εδρών. Είτε με λίστα, είτε ήμια ανοιχτά, είτε με, με ψήφο προτίμησης. Όλες αυτές οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση των εθνικών εκλογικών νόμων, κατά την άποψή μας, είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Η πρόταση για μια ευρωπαϊκή συνέλευση που θα συζητήσει αποκλειστικά αυτό το ζήτημα δεν είναι ακόμα όριμη κατά άποψή μας. Η Ευρώπη μόλις τώρα ολοκλήρωσε μια πολιτική μεταρρύθμιση και τα σημαντική και βιώνει αυτή τη στιγμή πολύ περίπλοκα προβλήματα οικονομικού κυρίως χαρακτήρα που δεν ε, κάνουν ε, δεν, δεν, δεν, θεωρούν ότι είναι, δεν επιτρέπουν να θεωρήσουμε καλό την ε, σύγκληση μιας συνέλευσης που αποκλειστικά αυτό το στόχο θα, έχω, θα έχει. Πιστεύουμε ότι Ε, μια συζήτηση τέτοια δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικό, οικονομικής κρίσης. Όντως, η Ευρώπη πολιτικά ε, πρέπει να κάνει μετα... Ε, συνέλευση για να κάνει συζητήσεις ευρύτερων θεμάτων, όχι μόνο τις εκλογές, περισσότερες ε, μεταρρυθμίσει. Για παράδειγμα, ε, για την οικονομική μεταρρύθμιση. Χθε η Τάσκο υπέβαλε έξι οδηγίε για τη μεταρρύθμιση τη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Τώρα δημιουργούμε το ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο για την επεξεργασία των, ευρω... των εθνικών προπολογισμών που πρέπει να διαμορφώνονται με την έγκριση της Κομισιόν, θίγοντας ή όχι την εθνική κυριαρχία. Όταν προκύπτουν όλα αυτά τα ζητήματα, ε, ίσως θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συζητηθεί ευρύτερα η προσαρμογή των συνθήκων στις νέες αυτές, στη νέα αυτή διακυβέρνηση. Αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο που θεωρούμε ως πολιτική ομάδα πως θα μπορούσε να επιτραπεί μια μεταρρύθμιση των συνθήκων και μια συνέλευση κατά συνέπεια. Τρίτον, δεχόμαστε το ότι είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση για ε, για τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια. Δεν έχουμε ωστόσο θετική άποψη σαν ομάδα για το ζήτημα αυτό και κάποιες άλλες παρατηρήσεις τηλεγραφικού χαρακτήρα. Πρώτον, φοβόμαστε ότι μπορεί ο κατάλογος, ε, το ψηφοδέλτιο αυτό να μην περιλαμβάνει, περιλαμβάνει όλων των χωρών και να δημιουργεί εθνική αντιπροσώπευση δυσανάλογη. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό, διότι Κάτι τέτοιο σε ορισμένε χώρε δεν θα γινόταν αποδεκτό. Μας ανησυχεί επίσης το γεγονός ότι ένας υπερεθνικό, ένα υπερεθνικό ψηφοδέλτιο θα δημιουργούσε δύο κατηγορίες βουλευτών. Βουλευτές Α ή Β κατηγορίες. Ε, επίσης υπάρχει ο κίνδυνο, ένα υπερεθνικό ψηφοδέλτιο να περιλαμβάνει τις μεγάλες προσωπικότητες ή κάποιες προσωπικότητες, μεγάλες ή μικρές δεν ξέρω, που είναι γνωστές στο δημόσιο, που είναι φημισμένες, χωρίς ωστόσο τούτο να συνδέεται πραγματικά με μια ουσιαστική κομματική αντιπροσώπευση. Μας ανησυχεί ε, το γεγονός ότι, μια, ότι ένα υπερεθνικό ψηφοδέλτιο θα είναι μακριά από τον πολίτη. Θα έχουμε δηλαδή δύο κάλπες ε, και στη δεύτερη κάλπη ο πολίτης θα ψηφίσει ανθρώπους που δεν ξέρει. Μας φοβίζει το ενδεχόμενο αποχής στο σημείο αυτό. Υπάρχουν λοιπόν επιφυλάξεις για το ζήτημα αυτό και θα ήθελα απλά να εκφράσω την ανησυχία μας για την πρόταση χωρίς να λάβω θέση ως ομάδα. Συμφωνούμε και τελειώνω πρόεδρε με τον στόχο της αύξησης της ε, συμμετοχής στις εκλογές των πολιτών. Μήπως ωστόσο θα έπρεπε να συζητήσουμε και άλλους τύπους και άλλες δυνατότητες. Για παράδειγμα, δεν θα ήταν σκόπιμο, μια και μιλάμε για τη μεταρρύθμιση όλων των πραγμάτων, να δούμε το ενδεχόμενο να υπάρχει υποψήφιος πρόεδρος της Επιτροπής σε κάθε, για κάθε πολιτική, μεγάλη πολιτική ομάδα. Δεν είναι αναγκαίο να προτείνουμε στους πολίτες την εκλογή ενός υποψηφίου ως πρόεδρο αναπολιτική ομάδα. Δεν θα ενίσχυε κάτι τέτοιο τα ευρωπαϊκά κόμματα ακριβώς. Περισσότερο και από αυτό το υπερεθνικό ψηφοδέλτιο. Δεν θα ενίσχυε η ιδέα την ιδέα μιας ευρωπαϊκή, ενός ευρωπαϊκού οικοδομήματος, το γεγονό ότι θα έχει έναν υποψήφιο πρόεδρο της Επιτροπή από του χριστιαδημοκράτες, από του σοσιαλιστέ, από του φιλελεύθερου, από του πράσινους. Μήπως θα μπορούσαμε να προτείνουμε ο πρόεδρος τη επιτροπή να προέρχεται από την ε, ε, πολιτική ομάδα που έλαβε τις ε, περισσότερε ψήφου. Θα θέλαμε να διευρύνουμε εν ολίγης την συζήτηση. Αναφέρω απλά αυτές τις επιφυλάξεις. Επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες ε, προς τον κύριο Νταφ που ε, έφεσε τη συζήτηση. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας και δεύτερο να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ε, ζητώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο προτάσεων από αυτές που περιλαμβάνει η έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Grazie a lei, come sempre chiarissimo. E πολύ ωραία, πολύ ωραία τα είπατε, ξεκάθαρα όπως πάντα και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Τόμας Κοκόφσκι που προέρχεται από την Πολωνία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το θέμα που συζητάμε συζητήθηκε ε, την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο της ε, Πολωνίας και ορισμένοι από τους ε, προλαλήσαντες είπανε ότι στην Πολωνία ούτε το Κοινοβούλιο ούτε και η κυβέρνηση έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος. Εγώ επιτρέψτε μου σύντομα να σας πω τι είπαμε στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι είναι πολύ καλή ιδέα ε, του να ε, παρουσιαστεί το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους ε, πολίτες. Βεβαίως εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και η συζήτηση ήταν αρκετά έντονη. Οι θέσεις λοιπόν που προτάθηκαν πρέπει να πω σε μεγάλο βαθμό δεν ήταν συμβατές και με τις θέσεις των μεμονωμένων πολιτικών κομμάτων. Όσον αφορά τώρα ε, στις εκλογικές περιφέρειες ε, και στο ημίκλειστο σύστημα, εμείς ε, στην Ολλανδία έχουμε ένα τέτοιο σύστημα για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Έχουμε 13 εκλογικές περιφέρειες για τις εκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό θεωρείται κάτι το θετικό τουλάχιστον η πλειοψηφία ε, αντιμετωπίζει θετικά την ύπαρξη αυτών των εκλογικών περιφερειών και έχουμε και ένα προτιμησιακό ή μη ανοιχτό ή μη κλειστό σύστημα όπως θέλετε να το χαρακτηρίσετε. Η ιδέα λοιπόν να υπάρχει μία ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια αυτή αντιμετωπίστηκε επιφυλακτικά. και μας θυμίζει την πολωνική, ε, τον πολωνικό εθνικό κατάλογο, τη λίστα που είχαμε κατά το παρελθόν. Και ελέγχθη κατά τη συζήτηση ότι μια τέτοια λίστα θα οδηγούσε σε ορισμούς ε, από τα κόμματα και δεν θα υπήρχε δυνατότητα επιλογής από πλευράς ε, πολιτών. Όπως είπαμε λοιπόν, ε, δεν θα υπήρχε δυνατότητα επιλογής, αλλά οι υποψήφοι θα ορίζονταν από τα κόμματα. Επίσης, μιλήσαμε και για την κατανομή των εδρών και όσον αφορά στην κατανομή των εδρών, νομίζω ότι είναι δύσκολο να περάσουμε αυτές τις αλλαγές στο Συμβούλιο. Όσον αφορά τώρα στην ε, εκλόγιμη ηλικία, το να έχουν δικαίωμα ψήφου και οι 16 ετής, αυτό είναι πολύ προχωρημένο. Αλλά ίσως ε, θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε το εκλογικό σύστημα. Αυτή η ιδέα ε, κρίθηκε θετικά και επίσης και η ιδέα αλλαγής της ημερομηνία, οι ευρωεκλογέ να γίνονται Μάιο. Και αυτό ε, κρίθηκε θετικά. Σας είπα λοιπόν, οι περισσότερες από αυτές τις απόψεις ε, αντιμετωπίστηκαν θετικά στο Κοινοβούλιο της ε, Πολωνίας και μόλις καταλήξουμε θα ανταποκριθούμε. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο. Άκουσες από τους περισσότερους από μας λόγια καλά γενικά, αν και υπήρξαν και κάποιες διαφοροποίησεις. Εγώ θα παίξω εδώ τον ρόλο του δικηγόρου του διαβόλου, γιατί υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με κάποιες από τις ιδέες σου. Και είτε στηρίζουμε τις ιδέες αυτές είτε όχι πρέπει να τις σχολιάσουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά. Όταν βλέπω πώς πηγαίνει η συζήτηση γύρω από τις ιδέες αυτές στα κράτη-μέλη, φοβάμαι ότι θα καταστεί αντιπαραγωγική σχετικά με την χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας και σχετικά με, τις, με, τους, με τα διαμεθοριακά ή διασύνοριακά ψηφοδέλτια. σε αυτή τη φάση δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς μια προεκλογική εκστρατεία κάτω από τη σημαία του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Όμως, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ορισμένα προβλήματα εφόσον προχωρήσουμε. Φαντάζεστε τον κίτρινο τύπο στη Μεγάλη Βρετανία λέγοντας ότι ο Άντζιου Νταφ στηρίζεται από χρήματα Ευρωπαίων Φεντεραλιστών που προέρχονται από την υπηρετική χώρα. Και φυσικά κάποιες συντηρητικές εκλογικές περιφέρειες στη χώρα σου μπορεί να έχουν πρόβλημα με αυτό και μπορεί να προκαλέσει κάποιες συζητήσεις εθνικιστικού τύπου ότι κάποιοι υποστηρίζονται από φρικτούς Ευρωπαίους φεντεραλιστές και αυτά όλα θα προκαλέσουν φοβίες περαιτέρω. Μπας περιπτώσει, εγώ δεν λέω ότι θα γίνουν όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι κάποιες από τις ιδέες σου μπορεί η συζήτηση γύρω από αυτές να είναι αντιπαραγωγική. Το δεύτερο θέμα, σχετικά με τα διασυνοριακά ψηφοδέλτια. πράγματι μπορεί θεωρητικά να γεννήσει μια πανευρωπαϊκή αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική και εξελίσσονται και οι εκλογές. Αλλά μπορεί όμως να δημιουργήσει και πολλά προβλήματα. Να σου δώσω ορισμένα παραδείγματα. Βλέπει κανείς από τη συζήτηση που προηγήθηκε τι ακριβώς πιστεύει ο κόσμος. Ξέρεις τι συζητήσεις γίνονται και στη δική σου χώρα, ε, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα ακολουθεί Σκέψου τώρα σε ένα ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο θα τσακώνεται ε, ο πολιτικός κόσμος ε, πόσοι θα είναι από τη μία χώρα, πόσοι θα είναι από την άλλη κτλ. Υπάρχει και το πρόβλημα του να μπορεί κανείς να είναι υποψήφιος σε δύο ψηφοδέλτια. Αν είσαι ένας ισχυρός πολιτικά θα τολμήσεις να μπεις μόνο στο διασυνοριακό ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι θα θέλουν οι πολιτικοί, όσο σημαντικοί και να είναι, να έχουν ένα δίκτυο ασφαλείας. Βάλτε με θα λένε στο διασυνοριακό, αλλά θέλω να είμαι και στο εθνικό ψηφοδέλτιο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η συζήτηση δεν είναι σοβαρή, γιατί όταν κάποιος είναι σε δύο ψηφοδέλτια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα προκαλέσει αρνητικά σχόλια. Ένα επιπλέον παράδειγμα. Αν ο πρόεδρος Μπούζεκ, λέμε τώρα θεωρητικά, είναι στο διασυνοριακό ψηφοδέλτιο και είναι και στο εθνικό ψηφοδέλτιο πριν από μένα. Τι κίνητο έχω εγώ. Θα υποστηρίξω την επιλογή φυσικά και ποιες θα είναι οι πιθανότητες να εκλεγώ εγώ. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας θα υποστηρίξει τον υποψήφιο της χώρας του για να ε, του δώσει την δυνατότητα να προωθηθεί και στο εθνικό ψηφοδέλτιο. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Και δεν θα είναι η επιλογή ας διαλέξουμε ένα από το εθνικό ψηφοδέλτιο και τον καλύτερο από το, ε, από το διασυνοριακό ε, ψηφοδέλτιο. Απλά θα διαλέγουν από το ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο αυτόν ο οποίος είναι από τη χώρα τους μόνο. Λοιπόν νομίζω ότι η ιδέα αυτή μπορεί να γελιοποιηθεί με λίγα λόγια γιατί θα αρχίσει να τσακώνεται ο κόσμο ποιος θα πάει μπροστά, πόσοι θα είναι από κάθε χώρα και σύν τη άλλη ποιον θα υποστηρίξει κανείς και για ποιους θα, λόγους θα τον υποστηρίξει και θα αναπαράγει στο ευρωψηφοδέλτιο τη λογική του εθνικού ψηφοδελτίου. Αυτά όλα πρέπει να τα σκεφτούμε σοβαρά. Δημιουργούν συγχύσεις. Αν κάθε πολιτικό κόμμα, σαν παράδειγμα, δημιουργήσει ένα ε, ψηφοδέλτιο 25 υποψηφίων, έτσι θα είναι. θα βάλουμε αλφαβητικά τον κόσμο που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο, θα τους ε, ιεραρχήσουμε. Ε, εν πάση περιπτώσει θα υπάρξουν ευρωπαϊκά ποσοστά εννοώ για ε, εκπροσώπους, για υποψηφίους εκτός της συγκεκριμένης χώρας ποιο θα είναι το ποσοστό τους. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο σε μια ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά μπορεί να γελιοποιηθούν διότι δεν θα τα έχουμε προπαρασκευάσει σωστά και οι εθνικιστικές αντιδράσεις θα είναι τέτοιες που θα εκμεταλλευτούν τις σωστές αυτές προτάσεις μόνο και μόνο επειδή δεν θα τις έχουμε καταθέσει καλά και δεν θα τις έχουμε εξηγήσει καλά. και τα πράγματα δεν θα πάνε έτσι όπως τα φαντάζεται αυτός που τα προτείνει. Λοιπόν, πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά, πρέπει να δούμε την αλληλεπίδραση που θα υπάρξει ανάμεσα στο εθνικό ψηφοδέλτιο και στο ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο. Ευχαριστώ κύριε Κογκλόφσκι το θέμα αυτού του εθνικού ψηφοδελτίου, επιτρέψτε μου να κάνω ένα μικρό σχόλιο, είναι μια σημαντική ιδέα. Και είναι και μια προσπάθεια να δώσουμε απάντηση στην απουσία ακριβώς των ευρωπαϊκών κομμάτων. Κόμματα τουλάχιστον που να λειτουργούν με τον ίδιο πολιτικό πολιτισμό και την ίδια αποτελεσματικότητα με τα εθνικά κόμματα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τον Άντριο Νταφ να διευκρινίσει αν σύμφωνα με τη δική του πρόταση οι επιπλέον 25 θα είναι πραγματικά επιπλέον ή θα ανήκουν στους πιθανώς 751. Υπάρχει και το πρόβλημα της πιθανής εναλλαγής των εθνικών αντιπροσωπιών Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ε, προβλήματα και λεπτομέρειες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει η λίστα η οποία κατατίθεται από το κόμμα και η λίστα αυτή μπορεί να αλλάξει πριν ε, τελικά ε, φτάσουμε στις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να δώσουμε βάρος και ουσία στο Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα. και αν περιοριστούμε στους 25 νομίζω ότι θα δημιουργηθούν κάποια επιπλέον πρακτικά προβλήματα. Ο κύριος Τηλιανίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς στο δικό μας κοινοβούλιο, στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, δεν έχουμε εξαντλήσει ακόμη τη συζήτηση για το θέμα Γι' αυτό οι πλήστες των απόψεων και προτάσεων που θα ακούσετε είναι περισσότερο προσωπικού χαρακτήρα και κομματικού. Ε, θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια στον κύριο Ντάφ εξ αρχής και μάλιστα όχι συγχαρητήρια τυπικού χαρακτήρα διότι πιστεύω ότι μέσα από αυτή την έκθεση παρόλο που υπάρχουν όντως ελλείψεις εν επιχειρεί να βάλει αυτό που λέμε στα ελληνικά το δάχτυλο επί των τύπων των ήλο Να πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα. Ε, δηλαδή να μπει στην ουσία. Που η ουσία για μας όλους εδώ που ασχολούμαστε χρόνια με την πολιτική είναι καταρχήν πως η κοινωνία θα συμμετέχει και θα μείνει κοντά στην πολιτική και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, η νεολαία της Ευρώπης θα νιώσει την Ευρώπη δική του. Μέχρι τώρα αποτύχαμε. Η μεγάλη αποχή των τελευταίων ευρωπαϊκών εκλογών έχει επιβεβαιώσει αυτή την αποτυχία και ας μην γελιόμαστε. Γι' αυτό, εάν μείνουμε κολλημένοι σε μια λογική ιδανικών λύσεων και ιδανικών εκλογικών συστημάτων, απλώς θα επιβεβαιώσουμε αυτό που λέει ο κόσμος ότι στην Ευρώπη απλώς συζητάμε γραφειοκρατικά όλη μέρα δίχως να επιχειρούμε λύσεις γρήγορες και ριζοσπαστικές. Και επειδή υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πρέπει να επιχειρήσουμε έστω για να έχουμε επιφυλάξεις. Και μάλιστα να γίνει σύντομα Γι' αυτό προσωπικά υποστηρίζω την ιδέα του Convention το συντομότερο για αυτό το θέμα, διότι όσο και αν δεν προσφέρει και θεωρείται συμπληρωματικό το εκλογικό σύστημα στη σχέση πολίτη και ευρωπαϊκών θεσμών, εν είναι αναφυσβήτητα το πρώτο βήμα. Επειδή η μεγάλη συζήτηση γίνεται για το πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο. Βασικά το Πανευρωπαϊκό Ψηφοδέλτιο τι επιδιώκει. Επιδιώκει να δημιουργήσει μια υπερεθνική αντίληψη των πραγμάτων και να την νομιμοποιήσει λαϊκά. Αυτό είναι το στίχημα και αυτός είναι ο στόχος. Άκουσα τις επιφυλάξεις του προηγούμενου συναδελφού, οι οποίες σε επίπεδο λεπτομεριών έχει δίκιο. Αλλά δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις. Όταν οι πλήστες των χωρών έχουν σε ό,τι αφορά τα, ψηφοδέλτια στις ευρωπαϊκές εκλογές λίστα. Γιατί να μην επιμείνουμε και οι προσωπικότητες οι οποίες είναι πολύ γνωστές πανευρωπαϊκά να μπαίνουν στο υπερεθνικό ψηφοδέλτιο και να δέχονται τη βάσανο της ψήφου ενώ να έχουμε λίστες στα ψηφοδέλτια σε επίπεδο εθνικό που σημαίνει οι λίστες υπάρχουν. Μπορούμε όλοι να γίνουμε συνήγοροι του διαβόλου και να βρούμε προβλήματα σε λεπτομέρειες. Η ουσία είναι να μην χάσουμε το στόχο. Και ο στόχος είναι η υπερεθνική αντίληψη των πραγμάτων και κυρίως ένα πανευρωπαϊκό όραμα σε επίπεδο καθημερινής πράξης, ειδικά στην εκλογική διαδικασία. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαμορφώσουμε αυτή τη λογική την πανευρωπαϊκή και είναι ένα πρώτο βήμα αυτό το οποίο θα πρέπει να στηρίξουμε ανεξαρτήτως ε, ε, συμπληρωματικών επιφυλάξεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που ρώτησε πριν ο Πρόεδρος, και έχει δίκιο, δεν πρέπει να αυξάνουμε έτσι εύκολα τους βουλευτές. Να φύγουμε από τους 751 γιατί δίνουμε την εντύπωση ότι δημιουργούμε θέσεις για τους εαυτούς μας. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, και λύνουμε πολλά από τα προβλήματα που έθεσε πριν ο, ο συναδελφός, είναι ότι από όποιες χώρες εκλεγούν ή του πανευρωπαϊκού ψηφοδελτίου να περιορίζεται ο αριθμός των ευρωβουλευτών στο εθνικό επίπεδο. Είναι μια λύση απλή που δεν ανατρέπει τις σημερινές ισορροπίες που υπάρχουν μεταξύ των αναλογιών των κρατών μελών. Και περιορίζει και την και το δίλημα που θα έχουν κάποιε προσωπικότητε σε ποια από τα ψηφοδέλτια θα μπουν ή πώ θα αντιδράσουν οι υποψήφοι, οι αθυποψήφοι του που θα είναι στα ψηφοδέλτια. Όμω θέλω να τελειώσω λέγοντα ότι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει επίσης είναι η, η αξιοπιστία, η απαξίωση που έχουν που έχει η λογική του κομματικού φαινομένου σήμερα και στον κόσμο και στην Ευρώπη, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπου η πολιτική αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα γιατί, γιατί ο πολίτης θεωρεί ότι δεν του έλυσε το μείζον πρόβλημα της προσωπικής του επιβίωσης. Και ακριβώς εδώ είναι που υπησέρχεται η σωστή άποψη του εισηγητή για το θέμα της, των ημιανοιχτών ληστών και της προτιμησιακής ψήφου. Ο πολίτης, κακά τα ψέματα, αναγνωρίζει στο πρόσωπο εξίσου σημαντικό ρόλο με το κόμμα. Και αν πέσουμε στην παγίδα ότι θα πρέπει να τον βάλουμε αποκλειστικά και μόνο στη λογική του κόμματος είτε του ευρωπαϊκού είτε του εθνικού, τότε κάνουμε μεγάλο λάθος. Θεωρεί ότι σήμερα που έχουν περιοριστεί πάρα πολύ οι ιδεολογικές διαφορές, και αυτό είναι θεωρώ κοινό τόπο, θα πρέπει όντω να αναδειχθεί και το πρόσωπο ω εξίσου σημαντικό στην εκπροσώπηση. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστούμε πολύ. Ε, κατ' ουσίαν ε, νομίζω, αν κατάλαβα καλά, ότι ε, προτιμάτε το να έχει κανείς το δικαίωμα ψήφου και εκτός των ληστών των κομμάτων που καταθέτουν τα κόμματα. Ο κύριος Ήλκεφ. Παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μου δημιουργείται η εντύπωση ότι έχουμε δύο διαφορετικές τάσεις. Έχουμε από τη μία αυτούς οι οποίοι έχουν ανθιβολίες και από την άλλη αυτούς οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ενθουσιασμό. Νομίζω ότι αυτή η διαφοροποίηση δείχνει ότι η έκθεση προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον και ότι εκ των πραγμάτων είναι μια έκθεση δυναμική, μια έκθεση σημαντική που θέλει να αλλάξει τα πράγματα, θέλει να αλλάξει ένα σύστημα το οποίο έχει λίγο ξεπεραστεί, ένα σύστημα το οποίο έχει παλιώσει πια, ένα σύστημα το οποίο έχει γεράσει θα έλεγα. Ο Άντζιου Νταφ μέσω της συγκεκριμένη έκθεσης απευθύνει ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Μας προκαλεί όλους να εκφραστούμε και να προσπαθήσουμε να χαράξουμε το σύνορο ανάμεσα στην πολιτική δεοντολογία από τη μία και στον πολιτικό πραγματισμό από την άλλη. Έχω την εντύπωση ότι η πρόταση του κυρίου Ντάφ σχετικά με την ύπαρξη 25 ξεχωριστών ε, υποψηφίων και κάνει την πρόταση αυτή για να ξεφύγουμε ακριβώς από την ε, πλευρά της πολιτικής πρακτικής η οποία μοιάζει περισσότερο με καζινό θα έλεγα και με φτηνού επίπεδου διαπραγματεύσεις. Ίσως εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι το καλύτερο μαθηματικό μοντέλο το οποίο, στο οποίο μπορούμε να προσφύγουμε για να δημιουργήσουμε αυτόν τον πανευρωπαϊκό εκλογικό χώρο που είναι το στόχο, ο στόχος του Άντριου Νταφ. Ταυτόχρονα ο Άντριου Νταφ λέγει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε κάποιες εκλογικές περιφέρειες, έστω και περιφερειακές σε μια πρώτη φάση και πάνω στις οποίες να βασιστούμε σε έφθετο χρόνο να προχωρήσουμε. Αυτό δεν ακούγεται σαν άσχημη ιδέα, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε ε, κάποιες περιφέρειες στην ουσία το μόνο που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε τις επιμέρους περιφερειακές διαμάχες που υπάρχουν στο εσωτερικό της κάθε χώρας και στην ουσία οι υποψήφοι θα είναι όμοιροι των ανταγωνισμών είτε σε εθνικό είτε και σε διεθνές επίπεδο εφόσον οι περιφέρειες αυτές έχουν προχωρήσει σε μια κάποια μορφή ολοκλήρωσης. Λοιπόν, η ιδέα αυτή της ευρωπαϊκής περιφέρειας δεν ακούγεται άσχημη. Τώρα το θέμα της ιδιότητας του πολίτη ή της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν βρίσκεται ε, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων τον τελευταίο καιρό. Σε ορισμένες χώρες στις οποίες έχουν υπάρξει κάποια βήματα σημαντικά προόδου σε ορισμένες χώρες ε, οι οποίες είναι και οικονομικά αναπτυγμένες υπάρχουν εκπρόσωποι άλλων χωρών λιγότερο αναπτυγμένων οικονομικά οι οποίοι αποτελούν αυτή τη στιγμή το 20-30% του πληθυσμού. Δεν πήγαν εκεί για να εκμεταλλευτούν το κοινωνικό σύστημα προστασίας, πήγαν εκεί για να δουλέψουν, γιατί η αγορά εργασίας τους είχε ανάγκη. Έχουμε λοιπόν ανάγκη και για διάφορους επιμέρους λόγους ένα ενιαίο εκλογικό σύστημα. Μια λύση φυσικά θα ήταν η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο μόνο στο μέλλον μπορεί να κρυφεί ουσιαστικά. Ας ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις όχι μόνο μαθηματικών και στατιστικών, αλλά ανθρώπων που έχουν εμπειρίες και ευαισθησίες σε σχέση με τη σύγκληση των συστημάτων, τη συνεργασία των συστημάτων και των ιδεών. Για να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπα στην αρχή σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβούλιων, των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Κάποια κοινοβούλια συζητάνε το θέμα αυτό επί της ουσίας, αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Είμαι βέβαιος ότι σε ορισμένα κοινοβούλια η συζήτηση που κάνουμε εδώ σήμερα είναι μια συζήτηση που πολύ απλά δεν έχει γίνει και θα γίνει με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση όταν γίνει. Αλλά θυμίζω ότι ήδη από το 2014 οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ήθελαν να έχουν στην διάθεσή τους κάποια νέα μέσα εκλογικά θα ήθελαν το εκλογικό σύστημα για τις ευρωεκλογέ να είναι καινοτόμο. Grazie alla parola eh, l'onorevole Gap. Ο κύριος Γκάψης από τη Λιθουανία παρακαλώ. Dėkoju labai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, tikrai įdomus pranešimas ir buvo... Αξιότιμε κύριε Σιγητά, κύριε Πρόεδρε, η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, όπως βέβαια και η όλη συζήτηση. Εγώ θα σας ε, παρουσιάσω τη δική μου την άποψη και όχι αυτή του κοινοβουλίου μας, γιατί σε εμά δεν έχει γίνει ακόμα συζήτηση για το θέμα αυτό. Έπεται βέβαια η συζήτηση. Σήμερα αν έπρεπε να αξιολογήσω την έκθεση αυτή, αν πράγματι αποτελεί επανάσταση ή όχι, κοιτάξτε, κάτω από το πρίσμα ενός πολιτικού θα έλεγα ότι πρόκειται για επανάσταση, γιατί ασχολούμεθα με θέματα που αφορούν όλους μας σε καθημερινή βάση, αφορούν ε, το αν θα εκλεγούμε ή όχι. Από την άλλη όμως, ε, ως ε, πολίτης ε, θα έλεγα ότι δεν είναι επανάσταση και μέχρι το 2014 ε, δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα. Τώρα, να πω και τα προσωπικά μου επιχειρήματα. Η Λιθουανία πολλές φορές ε, χρησιμοποιείται ως πείραμα, ως συνδικό χειρίδιο. Εμείς έχουμε διάφορα εκλογικά συστήματα. Το να προσθέσουμε 25 ή να έχουμε λίστες. Αυτό σε εμά δεν θα αλλάξει τίποτα. Για τους πολιτικούς μπορεί κάτι να αλλάξει, όχι όμως για τους πολίτες. Αμφιβάλλω αν ο Πρωθυπουργός μας ε, με βάση αυτό το, αυτή την πρόταση θα υποβάλει υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, παλιά είχαμε 13, τώρα εμεί θα έχουμε 12 ευρωβουλευτές. Γι' αυτό δεν έγινε καμιά μεγάλη πολιτική συζήτηση ε, και ούτε και άλλαξε πολύ ε, το πολιτικό σύστημα στη Λιθουανία. 12-13 αυτό δεν είναι και τόσο τραγικό και δεν επηρεάζει και την κοινή γνώμη. Αμφισβητώ μάλιστα το κατά πόσον αναλλάξει το σύστημα θα συνεπάγεται και σημαντικές αλλαγές στη Γερμανία, ακόμα και στην Ισπανία. Απλά όλα αυτά θα επηράσουν την πολιτική συζήτηση. Κατά νου πρέπει να έχουμε τους ε, εκλογείς. Ε, να δούμε τι ακριβώς επιθυμούν εκείνοι. Όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, τους ε, βουλευτές ε, πρέπει, ε, συγγνώμη, τους εκλογείς πρέπει να έχουμε κατά νου. Δεν θα πρέπει οι ευρωπαϊκές εκλογές να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης. Εξάλλου, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε και τον τρόπο εκλογής και την αλλαγή του, να γίνεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Γιατί με τον τρόπο αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να συμμετάσχει κανείς σε εκλογές. Εμείς μέχρι τώρα στην Λιθωνία δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να μπορεί κανείς να ψηφίσει ηλεκτρονικά, όμως στην Ισλανδία γίνεται κάτι τέτοιο. Η σημερινή συζήτηση ε, δεν εστιάζεται στον πολίτη. Ε, η συζήτηση είναι σημαντική για τους πολιτικούς αλλά όχι για τους ε, εκλογείς. Ανεξάρτητα τώρα κατά πόσον εκλογές θα γίνει το 2014 ή αργότερα, οι πολίτες δεν θα καταλάβουν τίποτα. Και με κάθε σεβασμό για τον εισηγητή, εγώ πιστεύω ότι αυτά που προτείνει είναι σημαντικά, όμως ε, ο πολίτης δεν θα καταλάβει τίποτα. Ε, και εμείς τον πολίτη πρέπει να έχουμε κατά νου τις ανάγκες του πολίτη και όχι των πολιτικών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μεσεσμίτ, ένας από τους αντιπροέδρους αυτής της Επιτροπής των Συνταγματικών Υποθέσεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνήθως μια τέτοια συζήτηση ε, μου προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα όταν εισαγωγικά την παρουσιάζει ο κύριος Ντάφη. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα, αλλά παρόλα αυτά η συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα. Η συζήτηση όμως που προηγήθηκε μέχρι τώρα είναι σχετικά απογοητευτική. Συμφωνούμε ότι υπάρχουν ε, ουσιαστικές δυσκολίες, αλλά υπάρχουν και ουσιαστικές ανάγκες για αλλαγές. Σε κάθε χώρα δεν υπάρχει δυνατότητα, σαν παράδειγμα, του να μπορεί να ψηφίζει κανείς με τον ίδιο τρόπο την ίδια κατηγορία υποψηφίων. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν διαφορές στα εκλογικά συστήματα, όλα αυτά θα πρέπει σε κάποια φάση να αλλάξουν. Και έχουμε και το γενικότερο ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο είναι η χαμηλή συμμετοχή. Τι συζητάμε όμως το σύνορα. Εμείς μιλάμε μόνο και μόνο για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος σε ένα σύστημα πιο ομοσπονδιακού χαρακτήρα, πιο φεντεραλιστικό. συζητάμε για κάτι το οποίο ποτέ δεν θα γίνει πραγματικότητα, έτσι εγώ νομίζω. Γιατί κανένα από τα εθνικά κράτη δεν θα δεχθεί ένα τέτοιο σύστημα. Γιατί χάνουμε το χρόνο μας λοιπόν και συζητάμε κάτι το οποίο ε, νομίζω ε, στο μυαλό του Ντάφ είναι ένα ωραίο όνειρο για το μέλλον. Ας μιλήσουμε για τα προβλήματα που έχουμε σήμερα και τι μπορούμε να κάνουμε για τα προβλήματα αυτά σήμερα. Συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα για να αυξηθεί το ποσοστό των πολιτών που συμμετέχουν στις εκλογές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ε, ότι θα το πετύχουμε με φεντεραλιστικές ιδέες και φεντεραλιστικές σε εισαγωγικά, το λέω αυτό, εκλογικές περιφέρειες στην Ευρώπη. Ο κόσμος δεν ψηφίζει και αυτό ισχύει για τη χώρα που εκπροσωπώ, είναι η έλλειψη πίστης και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον ρεαλισμό που θα πρέπει να χαρακτηρίζει αυτό εδώ το σώμα. Και νομίζω ότι η λογική που εξηγεί αυτή την απογοήτευση είναι σωστή και το μόνο που κάνουμε εδώ είναι να προσπαθήσουμε να προκαλέσουμε αύξηση του ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν εύκολο κύριε Ντάφ να πούμε σε όλους εκλογείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα για να εκπληρωθούν τα όνειρά τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να υπάρξει μεγαλύτερη ομοσπονδιακή Ευρώπη. Όταν θέσετε τις ιδέες σας στον κόσμο θα απογοητευτείτε βαθύτατα. Πρέπει αντίθετα να προτείνετε μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι τα βασικά εμπόδια για τη χαμηλή συμμετοχή, για τη μεγαλύτερη μάλλον υψηλότερη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές. Αυτά είναι θέματα τα οποία γνωρίζετε και τα έχετε αναφέρει, αλλά κανένας δεν τα συζητάει σε βάθος γιατί θέλετε να μιλάμε για ιδεολογίες και φιλοσοφίες και όχι για την πραγματικότητα. Λοιπόν, αγαπητέ Άντριου, πάρα πολύ συχνά ξεκινά ωραίε συζητήσει με οράματα για το μέλλον, αλλά καλό θα είναι να ασχοληθούμε και με τα καθημερινά προβλήματα. Η κυρία Παπαδημητρίου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθώ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα τελευταία 14 χρόνια από την έκθεση του Γιώργου του Αναστασόπουλου, τότε Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου μέχρι σήμερα και πιστεύω ότι είναι απόλυτα φυσικό και λογικό για το πόσο έχει καθυστερήσει και ενισχύω την άποψη του ΠΠΕ, του κόμματος που και υπηρετώ και του καθηγητή Σεφρίν ότι ίσως χρειάζεται ακόμα περισσότερος χρόνος. Πολύ καλή δουλειά έχει κάνει ο συνάδελφος ο κ. Ντάφα. Αλλά θα μείνω, μιλώντας για πιθανές παράγγελες απώλειες, στο σημείο 4 των προτάσεών του που ζητάει νομιμοποίηση, προτείνοντας την απευθεία συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, χωρίς τη μεσολάβηση των Εθνικών Κοινοβουλίων, παρά με ισχνό τρόπο. Πού θα μπουν τα εθνικά κοινοβούλια ουσιαστικά. Αποψής μου πρέπει να είναι παρόντα και εξάντε και ongoing, συνεχώς. Και συμφωνώ απόλυτα με τον τρίτο μιλητή από το Λουξεμβούργο σήμερα το πρωί που τόνισε ότι η αδιαφορία των Ευρωπαίων πολιτών από τις έως σήμερα διαδικασίες είναι ευθέως ανάλογη με την απουσία και την αμυδρή συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις δημοκρατικές ευρωπαϊκές διαδικασίες. Άκουσα τον Λόρδο Μπαούνες της Βουλής των Λόρδων, ο οποίος μάλιστα με τρόπο κατηγορηματικό είπε ότι οι εθνικοί βουλευτές δεν ενδιαφέρονται για να ενισχύσουν το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου. Διαφωνώ σε αυτό ως εθνική βουλευτής για 20 χρόνια και θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση. Σε όλα τα διακοινοβουλευτικά φόρα και σε όλες τις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών διεκδικεί περισσότερες ακόμα και ισότιμες αρμοδιότητες στο χώρο διάγραμμα της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής και για τα δύο όργανα και για το Ευρωκοινοβούλιο και για το σύνολο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πάντως, η διαφορά είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε εμείς οι εθνικοί βουλευτές οι απευθείας εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρόλου εκπροσώπου μας στις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κέντρο αβολοντέ χωρίς τη δική μας γνώμη την κοινά και διεξοδικά συζητηθήσα και συγκροτηθήσα. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι οι προβλέψεις της Λισαβόνας άρχισαν πάρα πολύ άσχημα υλοποιούμενες. Συμπερασματικά κύριε Πρόεδρε πιστεύω ότι το διακύβευμα για την απάντηση και τη σμίκρυνση του δημοκρατικού ελλείμματος είναι η άμεσα αναγκαίες για να συνοντηθούν, να συζητηθούν νέες ισότιμες και έντιμες σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλευτικού Κέντρου που μας φιλοξενεί σήμερα και της Κοινοβουλευτικής Περιφέρειας που συνιστούν τα Εθνικά Κοινοβουλιά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Παπαδημητρίου. Η παρέμβασή σας δείχνει τη σημασία και το βάρος που έχει αυτή η συζήτηση, όχι μόνο για το εκλογικό σύστημα, αλλά και για τις σχέσεις τις οποίες ε, πρέπει να έχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών σε σχέση με την πολιτική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Βέβαια δεν μπορούμε όλα να τα συζητήσουμε σε μία φάση, η διαδικασία είναι αυτή η οποία ξεκινάει. Danke, ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μπω στο ψητό και θα πω ότι ο κύριος Νταφ έχει δίκιο που λέει ε, με την η σκέψη β και γ ε, αναφέρεται και παραπέμπεται στο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να αναλάβει την πρωτοβουλία. Και η συζήτηση την οποία παρακολουθώ με ενδιαφέρον εδώ και αρκετή ώρα ε, με οδηγεί στο να διερωτηθώ μα πότε θα είναι κατάλληλη χρονική στιγμή. Μετά τις τελευταίες ευρωεκλογές ε, το Κοινοβούλιο, ε, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η Κυβερνήση έπρεπε όλοι από κοινού να ε, συναντηθούν και να δρομολογήσουν μια διαδικασία η οποία θα έχει να κάνει με τη φθήνουσα προσέλευση στις ευρωεκλογέ. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, αυτή η φθήνουσα συμμετοχή δεν αφορά μόνο τις ευρωεκλογέ, αφορά πάσης φύσεως εκλογές, περιφερειακές, εθνικές, αυτοδιοικητικές, οτιδήποτε. Εμένα λοιπόν ε, με απασχολεί το εξής. Αυτή την ε, έκφραση της δημοκρατικής τοποθέτησης των πολιτών. Πόσο σοβαρά την παίρνουμε, είτε πρόκειται για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είτε για το κράτος. Είτε, αν θέλετε, για την εκλογή ενός ε, δημάρχου, που είναι πολύ πιο απλό, γιατί εκεί ε, έχουμε να κάνουμε με τα καθημερινά του πολίτη. Το ερώτημα, λοιπόν, που πρέπει να μας απασχολήσει είναι κατά πόσον αυτή την ε, διτή συμμετοχή σε ευρωεκλογές και σε εθνικές εκλογές, πόσο σοβαρά την παίρνουμε σε σχέση με την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι Εθνικών Κοινοβουλίων λέω ότι πράγματι η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε στα κοινοβούλια ούτε στις πολιτικές ομάδες αλλά από ό,τι φαίνεται ούτε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχει καταλήξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και στη δική μου την πολιτική ομάδα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις. Θέλω λοιπόν να καταστήσω σαφές το εξής. Ε, εδώ είναι προσωπική μου βέβαια η άποψη. Τελικά τι θα κάνουμε με αυτήν την έκθεση. Βεβαίως η έκθεση ε, τα σωστά ερωτήματα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι με τα ερωτήματα που θίγει ο κ. Νταφ μπορούμε να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά και δεν λέω όπως είπε ο κ. Μέσσερ Σμίτ ότι όλα αυτά ε, απομακρύνουν ε, τα ενδιαφέροντά μας από τα πραγματικά προβλήματα του πολίτη. Εγώ λέω ότι αυτή η έκθεση είναι ένα καλό εργαλείο για να σκεφτούμε πώς μπορούμε να επιτρέψουμε τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Και βέβαια οι εκλογές είναι σημαντικό, αλλά όχι το μόνο εργαλείο. Επιτρέψτε μου να εκφράσω και κάποιες άλλες απόψεις που αφορούν σε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ελέγχθησαν για τα ευρωπαϊκά κόμματα. Νομίζω ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και αν είμαι σωστά ενημερωμένος, 10 είναι αυτά τον αριθμό, τα οποία αυτή τη στιγμή ε, παίρνουν από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Προπολογισμό περίπου 9 μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν είναι όμως ε, αυτόνομες ε, νομικές οντότητες. Έχουν αναγνωριστεί στο βελγικό δίκαιο λίγο πολύ. Άρα δηλαδή εμείς οι ίδιοι δεν αναγνωρίζουμε αυτά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Αυτά λοιπόν τα οποία μέχρι και το 2009 δεν είχαν το δικαίωμα να διεξάγουν προεκλογική εκστρατεία, πώς μπορούμε να περιμένουμε ότι αυτά θα επηρεάσουν την ε, διαμόρφωση βούλησης και συνείδησης ε, στον Ευρωπαίο πολίτη. Πώς μπορούμε να επιδιώξουμε να είναι αυτός ο διεισμός, δηλαδή ε, το εθνικό επίπεδο και το ευρωπαϊκό. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον κύριο Ντάφα ότι το θέμα δεν είναι να σκεφτούμε κατά πόσο μπορούμε να αποκτήσουμε άλλες 25 θέσεις, αλλά να σκεφτούμε ποια είναι η πολιτική ισορροπία ανάμεσα στα εθνικά και τα ευρωπαϊκά κόμματα. Ε, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, ε, σε τελική ανάλυση πρόκειται και για σκληρό ανταγωνισμό. Ποιο εθνικό κόμμα θέλει να παρετηθεί υπέρ ενός ευρωπαϊκού κόμματος. Αν είμαστε λοιπόν ειλικρινεί, το όλο θέμα αφορά ε, όχι μόνο τα κόμματα, αλλά και γενικότερα την πολιτική. Σε τελική ανάλυση ποια κυβέρνηση κράτους μέλους είναι πρόθυμη να εκχωρήσει κάποιες αρμοδιότητές της προς όφελος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Βλέπουμε λοιπόν ένα χάσμα ανάμεσα στην πολιτική συμμετοχή ε, τόσο της ε, αφρόκρεμας όσο και των ε, απλών πολιτών. Αυτό είναι το ένα μέρος. Και από το άλλο μέρος έχουμε τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το χάσμα πρέπει να γεφυρωθεί ως εκ τούτου θα πρέπει όλοι από κοινού να συμβάλλουμε στη μεταρρύθμιση ε, τη δημοκρατική αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Κατόπιν τούτου, εγώ προτείνω συγκεκριμένα το εξής. Να σκεφτούμε και να συζητήσουμε για το κατά πόσον αυτά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει και αυτά να ε, ορίζουν τους δικούς τους τους υποψήφιους. Όχι επιπρόσθετα, αλλά αναλογικά μέσα στον αριθμό που ήδη ισχύει. Διότι αυτά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, αυτά δεν εκφράζουν μόνο ε, τα δικά μας τα θέματα, αλλά προβάλλουν και τις δικές τους απόψεις, γιατί πιστεύουν αυτά για το μέλλον. Αυτή λοιπόν η διάσταση λείπει και κατ' με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το χάσμα ανάμεσα στη συνειδητοποίηση του πολίτη, τι δηλαδή γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πραγματικότητα. Θεωρώ ότι οι πολίτες ε, παρουσιάζουν εκλογική κόποση γιατί έχουν καταλήξει ότι και να κάνω τίποτα δεν γίνεται. Δηλαδή αν θέλετε οι πολίτες έχουν εξαντληθεί από την μη ικανοποιητική εξέταση των προβλημάτων του σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για ένα παράλληλο πρόβλημα και ε, πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε τόσο τα ευρωπαϊκά θέματα όσο και τα εθνικά. Ίσως λοιπόν η συνέλευση να είναι πραγματικά η σωστή λύση, η συνέλευση, η συγκέντρωση, πέστε το όπως θέλετε. Εκεί όμως να έχουμε εθνικούς, ε, ευρωπαϊκούς ε, βουλευτές, ευρωπαίους βουλευτές, ε, αλλά και κοινωνία των πολιτών και κυβερνήσεις, όλοι αυτοί να συγκεντρωθούν, διότι πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλα αυτά τα επίπεδα. Βεβαίως και είναι φιλόδοξος ο στόχος και εγώ δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι το 2014. Πρέπει όμως τώρα να επιληφθούμε του γιατι γιατί αλλιώς μετά από τρία-τέσσερα χρόνια θα είμαστε πάλι εδώ και θα λέμε α, ε, μειώθηκε περαιτέρω η προσέλευση στις εκλογές και θα έχουμε απλά κάνει μία τρύπα στο νερό. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, ε, για άλλη μια φορά ετέθη επιτάπητο στο νερο ευχαριστουμε λεει ο προεδρο για αλλη μια φορα ετεθη επιταπητο στο θεμα των ε, ευρωπαϊκών κομμάτων και ε, αναφέρθηκε επίσης και η σύγκρουση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα εθνικά και τα ευρωπαϊκά κόμματα. Και στο τέλος νομίζω ότι κατάλαβα και είναι εδώ ε, τρίτης ε, παραδοχής για να γίνουν πιο ευρωπαϊκές οι ευρωπαϊκές εκλογές. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Ντάφ, να έχουμε 25 θέσεις για, ένα, για μια ευρωπαϊκή λίστα. Τώρα αν κατάλαβα καλά, λέει ο πρόεδρος, εκφράστηκε και η άποψη του να ε, παρακρατηθεί ένα συγκεκριμένο, να προσημειωθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό για τα ε, ευρωπαϊκά κόμματα. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα δώσουμε το λόγο στον επόμενο ομιλητή, Γκοντίνα Νεάζη από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα, συνάδελφοι, πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχά ω νέο βουλευτή του Ουγγρικού Κοινοβουλίου ε, για την πρόσκλησή και να σα πω πόσο χαρά αισθάνομαι που με καλέσετε στη συνάντηση αυτή. Δύο εκπρόσωποι του Ουγγρικού Κοινοβουλίου έχουμε έρθει εδώ. Είμαι, τμήμα, είμαι μέρος, μέλος της ε, Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Σμιτ έφεσε ένα σημαντικό ζήτημα. Γιατί είναι τόσο επιφυλακτικοί οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η Επιτροπή μας στην Ουγγαρία δημιούργησε μία ε, υποεπιτροπή με την αρμοδιότητα την εξέταση και τη μελέτη της ε, παρεμβάσεις της αστυνομίας το 2006 μετά από ανώτερες ε, οδηγίες. Είναι λυπηρό βεβαίως αυτό που είχε συμβεί τότε. Κρίμα ιδίως διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεκίνησε να κάνει σχετικές έρευνες. Ο Επίτροπος Φρατίνη που ήταν ο αρμόδιος τότε δεν έκανε τίποτα σχετικά και δεν μέμφθηκε την, την Ουγγρική αστυνομία για τις ε, επεμβάσεις ε, της τότε. Λήφθηκαν τώρα χτες μια σειρά αποφάσεων για τη Γαλλία η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες και είναι πρόβλημα που γνωρίζουμε όλοι από δεκαετίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις σε πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Αυτό οδηγεί στις επιφυλάξεις των ψηφοφόρων. Η έκθεση DAF με βρίσκει σύμφωνο ως προς τη διάγνωση, αλλά τα υπόλοιπα μου δημιουργούν ερωτηματικά. Όντως υπάρχει αδιαφορία, υπά, όντως υπάρχει δυσφορία, όντως υπάρχει ε, απομάκρυνση. Ο κύριος Ντάφο τόσο μπερδεύει τα αίτια και τα αποτελέσματα. Ε, η Ευρώπη δεν μπορεί να δώσει σωστές, τις σωστές απαντήσεις σε μια σειρά ζητημάτων. Είναι, η Ευρώπη είναι ακόμα μοιρασμένη στις χώρες της Δύσης και τις χώρες της Ανατολής. Οι πρώην ε, κομμουνιστικές χώρες είναι χώρες που μόνο τυπικά έχουν τα ίσα, δικαιώματα με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Το ξέρει τι έγινε στην Ουγγαρία η κυρία Γκούρμα στο παρελθόν, ποιο είχε διατάξει την αστυνομία να πέμβει κατά των διαδηλώσεων. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα τυπικά. Επί τη ουσία, ωστόσο, το επίπεδο δικαιωμάτων σε κάποιες χώρες είναι τόσο χαμηλό που έχουν βαρεθεί οι πολίτες δεν προασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαντά σε ζητήματα όπως το γιατί μπόρεσε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα, μια χώρα όπως η Σλοβακία στην οποία ε, εφαρμόζονται ακόμα τα διατάγματα Μπένες και απαγορεύεται η αγορά και διώκονται Γερμανοί και Ούγγροι πολίτες. Εγώ συμφωνώ με όσους κατακρίνουν τις μεταρρυθμίσεις. Όχι τις μεταρρυθμίσεις αυτός καθεαυτές, ε, αλλά την ιδέα μεταρρυθμίσεων. Η πρόταση DAF δεν βλέπει το πρόβλημα από την οπτική γωνία του πολίτη. Πιστεύω ότι η λύση που πρέπει, αυτό που πρέπει να βρούμε είναι να δώσουμε μια ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος που μέσω του φεντεραλισμού, μέσω των ε, υπερεθνικών συνδυασμών που ε, πρέπει να επιβληθ, που, θέλουμε να επιβάλλουμε δεν νομίζω θα πετύχουμε να καλύψουμε το, το, το δημοκρατικό έλλειμμα. Τα εθνικά κράτη έχουν ρόλο, έστω και αν κάποιοι θέλουν να τον παραμερίσουν το ρόλο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια εικονική ε, πραγματικότητα. Ο κόσμος δεν θέλει περισσότερη Ευρώπη, θέλει, θέλει περισσότερη εθνική πραγματικότητα, εθνική βούληση. Όσο περισσότερο απομακρύνεται το εκλογικό σύστημα από τους πολίτες, τόσο λιγότερο οι πολίτες θα ενδιαφέρονται για την Ευρώπη. Πολλοί στην ευρωπαϊκή σημαία βλέπουν το μπλε, δεν βλέπουν τα αστέρια. Λίγες είναι οι υποσχέσεις που υλοποιούνται. Η Ευρώπη δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Να μιλήσω τώρα και για το θέμα των πολιτικών κομμάτων. είναι ένα ζήτημα που μου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά να σας πω την αλήθεια. Το σημείο 2β πιο συγκεκριμένα. Ξέρετε, εγώ είμαι νομικός. Και μπορώ να σα πω ότι όπως συχνά λένε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Η μεταρρύθμιση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή έχει στόχο, μάλλον ε, θα αποτύχει. Προορίζεται να αποτύχει. Οι προτάσεις αυτές θα έπρεπε να διατυπωθούν την ώρα που συζητούσαν τη που συζητούσαμε την συνθήκη τη Λισαβόνα. Και τότε είχαν συζητηθεί και απορρίφθηκαν. Εδώ τώρα δεν μιλάμε πια για συνθήκη τη Λισαβόνα, μιλάμε για κάτι καινούριο. Ζητήσαμε την άποψη του κόσμου. Θεωρεί ο κόσμο ότι αυτέ οι μεταρρυθμίσει είναι αναγκαίε. Πώ θα εφαρμοστούν. Πρόκειται λοιπόν εκ νέου για μια πρωτοβουλία που ξανά ξεκινά άσχετα και αδιά, ε, ε, άσχετα με τον πολίτη και διαφορώντα για τον πολίτη. Χωρί να ρωτάμε δηλαδή τι σκέφτεται ο πολίτη για τι προτάσει αυτέ. Λέτε εδώ Ευρωπαϊκή Αρχή, Ευρωπαϊκή Εκλογική Αρχή. Λέτε ε, ευρωπαϊκές, ε, ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκοί συνδυασμοί. όλα αυτά θα απομακρύνουν ακόμα περισσότερο τον πολίτη ο κόσμος θα βλέπει λίστες που δεν είναι εθνικές και θα το ακόμα περισσότερο από την Ευρώπη. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι προτάσεις αυτές είναι αντιδημοκρατικές. Το να συγκαλέσουμε τώρα μία συνέλευση είναι λάθος. Είναι λάθος ιδέα. Ευτυχώς η συνέλευση προηγούμενη δεν έδωσε αποτελέσματα συγκεκριμένα. Κα, κατέληξε σε αποτυχία όπως όλοι γνωρίζουμε. Πιστεύω ότι υπάρχει ήδη αρκετή γραφειοκρατία στην Ευρώπη και αυτό ακριβώς απομακρύνει τον κόσμο. Ο κόσμος νομίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν δουλεύουν για τον πολίτη και είναι ανησυχητικό το ότι διαπιστώνουμε πως συνεχίζονται, συνεχίζει να επιδιώκουμε χήμερες χωρίς να εμπλέκουμε τον πολίτη. Πάντως θεωρώ σημαντική τη συζήτηση και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Grazie per no. Σε ευχαριστώ για τα όχι σας σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ντάφ και στην Ευρώπη γενικότερα. Πράγματι αυτά που είπατε θα μας κάνουν να σκεφτούμε ακόμα περισσότερο. Στον εκπρόσωπο της ε, Πορτογαλικής Βουλής. Muito obrigado, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση την οποία έχει προετοιμάσει ο κύριος Νταφ δεν έχει ε, μελετηθεί επίσημα από την Πορτογαλική Εθνοσυνέλευση, ούτε και από το κόμμα μου, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Συνεπώς, οι απόψεις τις οποίες θα εκφράσω είναι ανεπίσημες και αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές μου θέσεις. Έχω την αίσθηση ότι η πρόταση του κυρίου Ντάφ είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια να δώσουμε μια πραγματική απάντηση στα προβλήματα τα οποία παρέθεσε ο κύριος Καζίνη στην προκαταρτική του εισαγωγή όταν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ότι οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ουσία κινδυνεύουν να θεωρηθούν δευτερεύουσες σε σχέση τουλάχιστον με τα εθνικά προβλήματα και τις, ε, και τα, τις εθνικές προκλήσεις στα πλαίσια των εκλογικών αναμετρήσεων. Όταν βλέπει κανείς την προοπτική του 2014, μιλάει για μια χρονική στιγμή η οποία είναι πάρα πολύ κοντά, οπότε ίσως δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί αλλά το ότι η προοπτική αυτή χρονικά είναι πάρα πολύ κοντά δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στα προβλήματα που έχουμε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να αποφασιστούν όπως το θέμα της ελάχιστης ηλικίας για συμμετοχή στις εκλογές, το θέμα των περιφερειακών διασυνοριακών εκλογικών περιφερειών, το θέμα του σεβασμού της, της ε, ε, μειούμενης ε, αναλογικότητας, όπως επίσης και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές απόψεις για, τις υπερεθνικές, για τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια ή τα διεθνικά αν θέλετε ψηφοδέλτια. Ε, κάποιοι υπερβάλλουν και θα μου επιτρέψετε να κάνω και εγώ το ίδιο Στην ουσία αυτό το οποίο αμφισβητείται είναι η, ακόμα και η δυνατότητα αυτών που θέλουν να πάρουν μέρος σε ένα φόρουμ το οποίο να αντικατοπτρίζει αυτό που είναι ιδανικό για ορισμένους σε σχέση με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Να υπογραμμίσω επίσης ότι η ιδέα ότι τα πολιτικά κόμματα μέχρι τώρα δεν έχουν ανταποκριθεί στην, στις προσδοκίες τις οποίες έχει ο πληθυσμός της Ευρώπης και η αίσθηση αυτή είναι συνέπεια του ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες έτσι ώστε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα το οποίο να προκαλέσει το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής κοινωνίας και να μην μείνει απλά αντικείμενο συζήτηση στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεπώς, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις προς ανατολισμού επί τη βάση ενός πολιτικού προγράμματος. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς την ενίσχυση της ιδέας του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος και οι προτάσεις του κυρίου Νταφ σε σχέση με τις εκλογικές περιφέρειες νομίζω ότι είναι αρκετά τεκμηριωμένες. Όσο για τον αριθμό των 25, ίσως θα πρέπει να δούμε αν ο αριθμός επαρκεί και αν μπορεί να αντιπροσωπεύσει σωστά τους λαούς και τους πολίτες της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει όμως ο αριθμός και η συζήτηση από τον αριθμό είναι ένα σημείο εκκίνησης μιας διαδικασίας η οποία θα προσδώσει κάποτε έναν πράγματι υπερεθνικό χαρακτήρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι τέτοιου είδους συνθήκες και χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δώσουν σάρκα και οστά και στο Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα και θα επιτρέψουν να αυξηθεί το επίπεδο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο πρόεδρος κύριος Λάινεν έχει το λόγο που ήταν και ο πρόεδρος πριν από μένα αυτής της Επιτροπής και τώρα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Παρακαλώ κύριε Λάινεν, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ο Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντο έχει τόσα πολλά θέματα να αντιμετωπίσει που συνήθω δεν έχει ευκαιρία να ασχοληθεί με αυτά που συζητούνται εδώ. Όμως αυτό το θέμα με ενδιαφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που είμαι Ευρωβουλευτής. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα ε, στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Θέμα επίσης που αφορά στην ε, εξέλιξη των ευρωεκλογών οι οποίες υπάρχουν με τη σειρά τους εδώ και 30 χρόνια. Κάθε φορά όμως ε, διαπιστώνουμε ότι η προσέλευση ακολουθεί φθήνουσα πορεία. Εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχω σε προεκλογικές εκστρατείες. Το 1990 πίστευα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και τότε πίστευα ότι αυτό οφείλεται στην εισαγωγή του ευρώ. Το 2004 εισήχθη το ευρώ, τα πράγματα πήγανε ακόμα χειρότερα και τότε ε, σκέφτηκα ότι οι άνθρωποι έχουν... Οι άνθρωποι φοβούνται το ευρώ, τουλάχιστον στη Γερμανία ήταν έτσι. Το 2009 είχαμε τη διεύνηση, τα πράγματα πήγαν ακόμα χειρότερα διότι διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς γιατί να πρέπει να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ. Και πράγματι τελικά δεν πρόκειται για ευρωεκλογέ. Τώρα έχουμε 27 διαφορετικές εθνικές εκλογές, 27 διαφορετικές προεκλογικές εκστρατείες και το δικό μου το κόμμα που είναι φιλοευρωπαϊκό ε, προσπάθησε κάθε φορά σε ευρωεκλογέ να αναδείξει ένα επίμαχο ε, ευρωπαϊκό πολιτικό θέμα. Ε, κάθε φορά όμως οι αντιπολιτεύσεις των κρατών μελών προσπαθούν σε ευρωεκλογέ να τις καταστήσουν λιδία λίθο για την εθνική τους κυβέρνηση. Και ό,τι και να λέμε, οι ευρωεκλογέ είναι αντικείμενο κακοποίησης από πλευράς ε, κυβερνήσεων και πολιτικών κομμάτων. Τα ευρωπαϊκά θέματα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Τα μέσα ενημέρωση ξέρουμε πώς λειτουργούν. Χρειάζονται γεγονότα, χρειάζονται ε, αγώνες ε, πολιτικής εξουσίας, ε, μάχες για απόκτηση εδρών και η, όλη η αντιπαράθεση δεν γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αντιπαράθεση παραμένει σε εθνικό επίπεδο. Εγώ λοιπόν το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η λογική συνέχεια από την ε, εισαγωγή των ευρωεκλογών το 70, κάτι το οποίο ήταν ένα μεγάλο θέμα τότε. Τότε υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις, ε, αρνητική αντιμετώπιση, αντίσταση. Ήταν ένα θέμα που χρειάστηκε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να οριμάσει στο πολιτικό σκηνικό μέχρι οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι δυνατόν απλά να στέλνει κανείς αντιπροσωπίες από τα Εθνικά Κοινοβουλία στο Στρασβούργο, γιατί τότε το Στρασβούργο έπαιζε. Ωραία ήταν όλα αυτά τη δεκαετία του 50 και του 60, αλλά αργότερα συνειδητοποίησαν ε, οι πολίτες και όλοι οι άμεσα εθνείς... ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τώρα λοιπόν, μετά από 30 χρόνια, φτάσαμε σε μια χρονική στιγμή που πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Οι ευρωεκλογέ να γίνουν πραγματικά ευρωπαϊκές εκλογές. Εγώ ήμουν εισηγητή στο Κοινοβούλιο για το καταστατικό των ευρωπαϊκών κομμάτων. Το 2004, λίγο πριν από τις ε, ευρωεκλογές, κατέστη δυνατόν κάτι τέτοιο και πρέπει να ομολογήσω το οφείλουμε στην ελληνική προεδρία. Η ελληνική προεδρία τότε είχε ε, την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί είχαν επιφυλάξεις στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στο Λουξεμβούργο και νομίζω και στο Βέλγιο, αλλά και στην Ελλάδα είχαμε την εξής κατάσταση. Ε, τα κόμματα δεν μπορούσαν να δεχθούν ε, ενίσχυση από ιδιώτες και από εταιρείε. Αυτό όμως γίνεται σε άλλες χώρες. Και πώς μπορεί να εξευρεθεί μία λύση και επειδή η Ελλάδα δήλωσε αποχή, πέρασε τελικά αυτή η δυνατότητα. Ε, προέκυψε λοιπόν το καταστατικό των ευρωπαϊκών κομμάτων. Κάτι έγινε, όμως τα κόμματα δεν μπορούν να δουλέψουν. Τι να κάνουνε. Δεν είναι λέσχοι, ρόταροι ή οτιδήποτε άλλο, τα κόμματα θέλουν εξουσία. Θέλουν σε εκλογές να αποκτήσουν έδρες για να έχουν μεγαλύτερη εξουσία. Τα ευρωπαϊκά κόμματα όμω δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ούτε καν ένα καλό προεκλογικό ευρωπαϊκό αγώνα δεν μπορούν να διεξάγουν. Γι' αυτό λοιπόν ποτέ δεν θα γίνει τίποτα αν και τα ευρωπαϊκά κόμματα δεν μπορούν να διεκδικήσουν έδρες και αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Είχαμε την έκθεση του κυρίου Αναστασόπουλου ήδη κατά τη δεκαετία του 90. Τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε το 10% των εδρών να ορίζεται από ευρωπαϊκές ε, λίστες. Ο κύριος Ντάφ είναι πολύ μετριοπαθής και λέει 27. Ε, τώρα το Κοινοβούλιο μεγάλωσε και ζητάμε κάτω από το 10%. Ακούω λοιπόν από όλους τα ίδια επιχειρήματα που ε, αγνωρίζω με παρηγορεί το ότι ο κύριος ε, Μάλλον, ο κύριος Φαγιό λέει συνέχεια τα ίδια. Εγώ είμαι γείτονά του, είμαι ακριβώς στην ε, διπλανή περιοχή. Ακούω λοιπόν την άποψη να έχουμε μία λίστα που να είναι λίγο διασυνοριακή, να αφορά όμορες περιφέρειες. Αυτό όμως δεν είναι ευρωπαϊκό ε, απευθύνομαι σε σένα. Οι πολίτες δεν θέλουν ε, μια λίστα που να αφορά την περιοχή του Ζαρ, ε, το Λουξεμβούργο και μια άλλη περιοχή της Γερμανίας. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ζούμε σε μια εποχή των μέσων ενημέρωση, όλα παίζουν μέσα από το διαδίκτυο και όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία, τα μέσα ενημέρωση αυτομάτως ε, θα έφτιαχναν μια πλατφόρμα για συζητήσεις. Και ναι μεν στην Ευρώπη ζούμε σε μία βαβυλώνα με τη διερμηνία, το πράγμα όμως λειτουργεί, γίνεται με τον τρόπο αυτό. Και έτσι θα αποκτούσαμε μία τελείως διαφορετική δυναμική στην ευρωπαϊκή συζήτηση και στους πολίτες που θα είχε νόημα, που θα παρουσίαζε με νόημα τις ευρωεκλογέ. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έφτασε η χρονική στιγμή οι πολίτες να έχουν δύο ψήφους στις ευρωεκλογέ. Μία ψήφο, όπως μέχρι τώρα, για, την, τον εθνικό για τις εθνικές λίστες, σε μεγάλες χώρες έχουν και περιφερειακές λίστες. Εκεί τέλος πάντων να μην αλλάξει τίποτα, εμείς να μην παρέμβουμε, όμως λείπει ε, ο άλλος βραχίωνας, η άλλη πλευρά. Αυτή, αυτό το στοιχείο της ε, αμυγούς ευρωπαϊκής λίστας. Κάτι τέτοιο λοιπόν ε, θα αντικαθρέφτιζε και την νομιμοποίηση, την ευρωπαϊκή νομιμοποίηση των κομμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση κρατών και είναι ένωση πολιτών. Από την συνθήκη του Μάστριχτ έχουμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και απλά αυτή ε, δεν λειτουργεί, ε, δεν έχει προχωρήσει. Από το 90 δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου, δηλαδή εδώ και 20 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω αν γίνεται, βέβαια το 2004 είναι πολύ κοντά για να είναι ε, φυκτό, ας γίνει το 19 τέλος πάντων πρέπει όμως να πιστούμε για το θέμα και να λέμε ότι θα είναι υποψήφιοι που θα είναι πολύ μακριά από τους πολίτες, δεν γίνονται αυτά εγώ ζω σε μια μεγάλη χώρα με 82 εκατομμύρια και όλοι οι υποψήφοι είναι και μακριά μας αλλά και πολύ κοντά μας, πολύ κοντά μας γιατί ε, τους δείχνουν συνέχεια τα μέσα ενημέρωσης, ε, βλέπουμε τα πρόσωπά τους ε, στις ε, ευρωλίστες οι άνθρωποι θα ήταν γνωστοί στη χώρα τους και μέσα από τα μέσα ενημέρωση και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, έτσι λοιπόν αυτά που παρουσιάζει ο κύριος Νταφ είναι πολύ φιλόδοξα, ίσως υπερβολικά φιλόδοξα. Εγώ θα να από πάρα πολλές λεπτομέρειες αυτά που γράφεις, Άντριου. Αυτά είναι όλα καθαρά τεχνικής φύσεως. Ε, μπορούμε να τα καταργήσουμε. Γιατί το κομβικό στοιχείο είναι η τομή, μια τομή όπου παράλληλα με τις εθνικές να έχουμε και ευρωλίστες για να έχουμε ευρωσυζήτηση και να ελοπίσουμε την ευρωδημοκρατία. Προφανώς χρειαζόμαστε αλλαγή της συνθήκης. Ε, το καλύτερο θα ήταν μέσω συνέλευσης, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Έχουμε, ας πούμε, την ενταξιακή συνθήκη της Κροατίας. Θα έχουμε και μια επόμενη ενταξιακή συνθήκη. Θα υπάρξουν πολλές δυνατότητες όπου το θέμα αυτό μπορούμε να το θέσουμε επιτάπητος. Τελευταίο μου σημείο όσον αφορά αυτή την τομή που θα ήταν ε, διαρθρωτική τομή. Προφανώς και θα υπάρξουν πολλές αντιδράσεις. Θα είναι οι εχθροί της Ευρώπης που δεν θα θέλουν αυτή τη λύση. Θα έχουμε τους ευρωσκεπτικιστές που λένε κάτι τέτοια δεν γίνονται και αυτοί θα είναι ε, ενάντι. Αλλά η... τα εθνικά κόμματα και αυτά το, τα, η καθεστική ετάξη των ε, κομμάτων και αυτοί θα διαφωνήσουν. Όπως σας είπα, εγώ επεξεργάστηκα το καθεστικό των ευρωπαϊκών κομμάτων και τώρα με την πρώτη αναθέωση τι κάναμε, ε, προβλέψαμε και ευρωπαϊκά ιδρύματα. Η δική μου πολιτική οικογένεια έχει ευρωπαϊκά ιδρύματα. Στη Γερμανία έχουμε πολύ ισχυρά ιδρύματα, το Konrad Adenauer, ε, το Friedrich Ebert, ε, ο Μπέλ και πολλοί άλλοι στη Γερμανία έχουν ιδρύματα. Ε, όμως δεν έχουμε ευρωπαϊκά ιδρύματα. Αλλά τι το εξή ερώτημα. Γιατί να υπάρχουν αυτά τα ιδρύματα. Τέλος πάντων, εδώ και δύο χρόνια υπάρχουν, καλά τα πάνε, έγιναν και κάπως γνωστά. Έτσι θα γίνει και εδώ. Θα έχουμε πάρα πολλούς που θα έρθουν και θα μας ε, βομβαρδίσουν ε, γιατί δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί όλα πάνε καλά. Όχι, δεν βαίνουν όλο καλώς. Οι ευρωεκλογέ επιδεινώνονται συνεχώς. Και στο φίλο από την Ουγγαρία μπορώ να πω, ίσως ε, γι' αυτό να φταίει η κακή πολιτική, μπορεί όμως και όχι. Η δημοκρατία στη τελική ανάλυση είναι δούνε και λαβίν. Εμείς επιθυμούμε καλύτερη δημοκρατία η συζήτηση όμως δεν γίνεται. Μα πού γίνονται ευρώ Τρει ε, Τρεις εβδομάδες πριν από τι ευρωεκλογέ. Αλλιώ καμία συζήτηση για την Ευρώπη ίσως να γίνεται μια συζήτηση όταν έχουμε κάποιο σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώ τίποτα δεν κουβεντιέται. Βλέπετε λοιπόν πόσο παθιασμένο είμαι. Εδώ και 15 χρόνια ε, ασχολούμαι με το θέμα και θα έλεγα, Άντριου, όταν θα ψηφιστεί η έκθεσή σου, να παρετηθεί από κάποιε λεπτομέρειε που θα μπορούσαν να θίξουν ευρωπαϊκά συντάγματα και ευρωπαϊκέ ε, ή εθνικέ νοοτροπίε. Εθνικά συντάγματα και εθνικέ ε, νοοτροπίε. Το κομβικό ε, σημείο είναι οι ευρωλίστες και ε, για τις λεπτομέρειες ε, μπορούμε να συζητήσουμε είτε στη διακυβερνητική ή αν τα πράγματα πάνε, πάνε πάρα πολύ καλά στο πλαίσιο μιας συνέλευσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Λάινεν. Ο συνάδελφος κύριος Βιάλα από τη Γαλλική Γερουσία έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την ε, σημερινή μας συντάντηση και ευχαριστώ τον κύριο Ντάφ για την παρουσίασή του και για τα τεχνικά ζητήματα για να απαντήσω στον τελευταίο μιλητή που φαίνεται ότι θεωρεί πως τα τεχνικά ζητήματα πρέπει να τεθούν κατά μέρου. Πρώτο θέμα για το χρονοδιάγραμμα. Δεν γνωρίζω αν η Ευρώπη θα είναι έτοιμη για το 2014 με τις αλλαγές αυτές. Σας συγχαίρω όσο που ξεκινήσατε ήδη από σήμερα τη συζήτηση αυτή, διότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Να σας πω ότι και η Γαλλική Γερουσία αποφάσισε πρόσφατα να συζητήσει το θέμα αυτό της εθνικής εκλογικής περιφέρειας. Είναι μια συζήτηση που λαμβάνει χώρα μόνο στη Γερουσία βεβαίως. Πρέπει να λάβει θέση και, το, ε, και η Εθνοσυνέλευση. Δείχνει όμως ότι τις ίδιες, ε, τους ίδιους προβληματισμούς έχουμε. Κάποιες παρατηρήσεις για αυτά που είπε ο κύριος Νταφ καταρχάς. Καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε ότι η ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία είναι πολύ πιο θεμελιώδης και πρέπει να μην θεωρηθεί ότι είναι τεχνικό κατά βάση ζήτημα, γιατί μιλάμε για την καρδιά της ενίσχυσης της δημοκρατίας, το κέντρο της ενίσχυσης της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αγαπητοί συνάδελφοι, μην κρυβόμαστε. Οι πολίτες, και αυτό το ενισχύει η κρίση, έχουν πολλά ε, ερωτηματικά εναντί της Ευρώπης. Μπροστά στην η ενίσχυση αυτή της Ευρώπης πρέπει να συνοδεύεται ταυτόχρονα με το σεβασμό των ταυτοτήτων, των συλλογικών ή τοπικών ταυτοτήτων. Νομίζω ότι την Ευρώπη τη μαθαίνει κανείς καλύτερα όταν δουλεύει για τη σχέση της Ευρώπης με τα έθνη κράτη και με τις περιφερειακές δομές. Να, υπο... να μπω και σε κάποια τεχνικά, είπα κάποια τεχνικά ζητήματα και μετά θα μπω και σε κάποια πολιτικά. Τεχνικά πρώτα. Για το ζήτημα των ε, ασυλιών και των προνομίων των ευρωβουλευτών. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι τελείως ε, έξω από τις εθνικές συζητήσεις με του συναδέλφους ε, στη Γαλλική Γερουσία μετέχουμε εδώ και λίγους μήνες σε μια επιτροπή που έχει συσταθεί για να χτενίσει τρόπον τεινά το θέμα των εκλογών σε εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο. Είναι δύσκολο να υιοθετούνται κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να συσχετίζονται με το τι γίνεται σε εθνικό πλαίσιο. Το θέμα της, εκλογική της εκλογικής ηλικίας 16-18 δεν είναι μόνο πολιτικό. Πώς μπορούμε να μιλούμε για κάτι τέτοιο χωρίς να υπάρχει εναρμόνιση της ε, ηλικίας ε, ε, της, για οποία κάποιος έχει το δικαίωμα ψήφου σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που σχετίζεται με μια σειρά παρα, παρεμφερών δικαίων. Η η νομική ενηλικίωση, για παράδειγμα, ε, δεν, μπαίνουν, δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε τέτοια ζητήματα ελαφρά την καρδία. Τρίτο ζήτημα, χωρί να θέλω να δείξω ότι θέλω να περιορίσω τη συζήτηση σε τεχνικά ζητήματα, έστω και φταίνει σε θεμελιώδη. Η κατάσταση των ε, πολιτών άλλων χωρών που κατοικούν σε άλλη χώρα της Ένωσης. Τέσσερα εκατομμύρια είπατε είναι στην Ευρώπη αυτή. Αναφέρθηκε η ειδική κατάσταση στο Λουξεμβούργο. Καλό θα ήταν από καιρού εις να βλέπουμε τις ακραίες περιπτώσεις. Σύμφερα, σήμερα το ζήτημα αυτό εμφανίζεται με την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ε, αλλοδαπών πολιτών της Ένωσης. Δεύτερο μεγάλο Δεύτερη ομάδα, μεγάλη ομάδα παρατηρήσεων πολιτικού χαρακτήρα. Η πρόταση για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας. Το θέμα του αριθμού των μελών αναφέρθηκε, δεν θα αναφερθώ ξανά. όπως σωστά είπε ο κ. Νταφ, ε, το θέμα του εκλογικού τύπου θα, θα λυθεί από τους μαθηματικούς. Φαντάζομαι ότι τα κόμματα θα έχουν μια κοινή προσέγγιση στο θέμα αυτό. Από την άλλη πλευρά, αυτά που είπατε εσείς πρόεδρε, όταν είπατε ότι η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να τραβήξει μεγάλες ευρωπαϊκές προσωπικότητες στην προεκλογική εκστρατεία. Εδώ είναι το βασικό ερώτημα του τι περιμένουμε από αυτή την πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια. Το λέω πολύ απλά. Η Ευρώπη συχνά αντιμετωπίζει τη μομφή ότι κρύβει πολιτικές ε, επιθυμίες πίσω από τεχνικά ζητήματα. Η πανευρωπαϊκή αυτή εκλογική περιφέρεια πρέπει να τεθεί με πολύ σαφή τρόπο. Τι θέλουμε από αυτή την εκλογική περιφέρεια, να εξισορροπήσουμε την αντιπροσώπευση, να αναδείξουμε μια νέα γενιά ευρωβουλευτών που θα είναι Ευρωπαίοι ομοσπονδιακοί βουλευτές και όχι ε, εθνικοί ευρωβουλευτές. Νομίζω ότι το σημείο αυτό θα έπρεπε να το δούμε πιο προσεκτικά. Δεν είναι ένα παρεμπίπτον, αλλά θεμελιώδες ζήτημα. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο αναφερόμενο σε αυτά τα λίγα σημεία θα παρέπεμπα, θα μιλήσω τώρα για την πρόταση μιας θεματικής συνέλευσης. Η εκλογική ευρωπαϊκή διαδικασία, πιστεύω, περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά ζητήματα. Κάποια μπορεί να φαίνονται τεχνικά, αλλά πίσω από τα τεχνικά κρύβονται πολιτικές ισχυρές προσδοκίες και που ούτως ή άλλως δεν αφορούν αποκλειστικά την Ευρώπη, αλλά και την ζωή των εθνικών θεσμικών δομών, κρατών τοπικής αυτοδιοίκησης. Και γι' αυτό το λόγο, κλείνοντας και ευχαριστώντας εκ νέου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργάνωσε τη συνάντηση αυτή, θα ήθελα αυτή η θεματική συνέλευση να επιτρέψει μια πιο διεξοδική ανάλυση όλων αυτών των ζητημάτων που είναι στο κέντρο των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρόνς έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δημοκρατία είναι κάτι του οποίου ηγείται ο λαός, όχι μια φθαίρετη δράκα ανθρώπων. Το Βέλγιο έχει την τύχη να έχει δύο βέβαια, ίσως και τρεις λαούς, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως κάποτε να υπάρξει ευρωπαϊκή ταυτότητα που θα αντικαταστήσει την εθνική ταυτότητα. Ο κύριος Ντάρ θα κάνει ό,τι μπορεί, όχι εγώ. Δεν έχει συμβεί όμως κάτι τέτοιο ακόμα. Αν αυτή η ευρωπαϊκή ταυτότητα πράγματι αναπτυχθεί, τότε ίσως θα ήταν καλό να προχωρήσει κανείς σε πανευρωπαϊκές εκλογικές περιφέρειες. Αλλά αν δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή ταυτότητα κάτι τέτοιο θα ήταν άχρηστο. Νομίζω ότι η συνταγματική αλλαγή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που υπάρχουν σε επίπεδο ταυτότητας και όχι να προσπαθεί να τις ε, δημιουργήσει. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον του κοινού για την ε, διευρωπαϊκή αυτή εκλογική περιφέρεια. Και τα κόμματα τα οποία είναι εναντίον αυτών των αντιλήψεων, αν δείτε την παράγραφο 2β και την τροπολογία 5, θα δείτε ότι τέτοιου είδους κόμματα θα ε, αποκλειστούν. Οι 25 έδρες στην ουσία θα είναι ένα δώρο στην ευρωπαϊκή πολιτική τάξη εις βάρος αυτών που έχουν εθνικές αντιλήψεις. Οι 25 αυτές είναι επιπλέον υποτίθεται, αλλά όσο θα αυξάνεται ο αριθμός ε, των ε, βουλευτών, δεν θα αυξάνεται και ο αριθμός αυτών που θα εκλέγονται με το ενίο ψηφολόγιο. Ε, και στο τέλος λοιπόν στην ουσία θα λειτουργούν αυτοί οι 25 εις βάρος των άμεσα εκλεγμένων οι εκλογικές περιφέρειες θα γίνονται μικρότερες και απλά θα καλύπτονται τα έξοδα των μεγάλων κομμάτων. Τώρα, για την δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις αυτών που κατοικούν σε μια χώρα. Δεν θα πρέπει να του στερείται το δικαίωμα αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να ασκούν το δικαίωμα αυτό στην χώρα στην οποία ζουν, αλλά στην χώρα προέλευσης με ταχυδρομικό τρόπο ή με κάποιον άλλο. Μάγερ από την Αυστρία. είμαι πρόεδρε, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είχα μέχρι τώρα ασχοληθεί με την έκθεση. Ε, θα κάνω όμως κάποιες ε, παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι η έκθεση DAF αποτελεί μια πολύ καλή βάση για συζήτηση και δεν θα ήθελα, όπως την άλφος ε, κύριος Μέστα Σμίτ και ο κύριος Γκάντινοτς, ε, να καταδικάσω ε, την έκθεση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία για συζήτηση στην έκθεση αυτή και όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά κυρίως στα Εθνικά Κοινοβούλια. Νομίζω ότι η έκθεση περιλαμβάνει κάποια πολύ καλά στοιχεία. Ελέγχθησαν πάρα πολλά ή αν θέλετε λέχθησαν όλα. Εγώ όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια σημεία, κυρίως όσον αφορά το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Θα ήθελα να υπερασπιστώ τους νέους, γιατί εμείς ε, στην ε, Αυστρία ε, είχαμε μια τέτοια μακρά συζήτηση. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στους νέους. Οι νέοι σε ηλικία 16 ετών είναι ενήλικες και μπορούν να πηγαίνουν στις κάλπες ε, να ψηφίζουν. Αυτή η υπερεθνική ευρωπαϊκή λίστα με τους 25 και διερωτώ με γιατί 25 και όχι 27 ή αν ε, έχουμε διεύνηση, γιατί να μην έχουμε έναν άλλο αριθμό με βάση τη διεύνηση. Το 25 δεν το καταλαβαίνω καλά. Βέβαια θεωρώ ότι είναι ένα επιπρόσθετο δημοκρατικό εργαλείο, το 25. Και η ευρωπαϊκή λίστα θα πρέπει να συστηθεί και κάτω από αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση. Βεβαίως το θέμα που τίθεται είναι ε, πώς ε, θα παρουσιάζονται οι υποψήφοι. Ε, θα μπορούν να είναι και ευρωβουλευτές και εθνικοί βουλευτές. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον συζητήθηκε και κάτι άλλο που εγώ θέλω επίσης να το υποστηρίξω. Εν τω μεταξύ, σε πολλές χώρες έχουμε πρόβλημα με το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ενισχυθεί αυτό. Όπως άκουσα σήμερα, πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρώπη γιατί κάτι τέτοιο ε, θα έχει θετική επίχυση στα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με αυτό που ελέγχθη από τον κύριο Λάινεν, από, ότι από τον 90 έχουμε επιδείνωση της κατάστασης ε, και διερωτώ με το 2014 τι θα γίνει τελικά. Φοβάμαι μήπως δεν πάει κανείς να ψηφίσει και αυτό θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ίσως λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επανέλθουμε με τον τρόπο αυτό σε μια ικανοποιητική προσέλευση, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις εκάστοτε εθνικές εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μενσαμάρετ από την Εσθονία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Στη Βουλή της Εστονίας δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το θέμα αυτό και προβλέπεται να γίνει η συζήτηση για την πρωτοβουλία των πολιτών σήμερα το απόγευμα. Άκουσα πολύ προσεκτικά του συναδέλφου μου και βλέπω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε οι ευρωεκλογές να οργανωθούν σωστότερα και να υπάρξει και μεγαλύτερη συμμετοχή. Στην Εσθονία μπορεί ο κόσμος να ψηφίζει ηλεκτρονικά με την ταυτότητά τους και η συμμετοχή στις εκλογές το 2009 ήταν ικανοποιητική. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος είναι σχετικά απογοητευμένος γιατί στις ευρωεκλογές, ναι μεν μιλάμε για ευρωπαϊκού υποτίθεται ενδιαφέροντος εκλογές, αλλά τα κόμματα χρησιμοποιούν τις εκλογές αυτές για να λύσουν τα προσωπικά τους, εννοώ τα, τα κομματικά τους προβλήματα. και δημιουργείται και σύγχυση στον κόσμο γιατί και το, κόσμο, το κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανήκουν και τα δύο στην φιλελεύθερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πράσινοι προσπάθησαν να κατέβουν με μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα αλλά τα μέσα ενημέρωσης της Εστονίας αδιαφόρησαν πλήρως για τους Εστονούς πρασίνους Υπήρξε συζήτηση σε σχέση με κοινωνικά θέματα όπως η υποστήριξη ε, των οικογενειών Έτσι και αλλιώ τα κόμματα κατέβηκαν με συγκεκριμένη λίστα προκαθορισμένη, οπότε δεν υπήρχε η δυνατότητα ουσιαστικά για τον κόσμο να διαλέξει. και ο κόσμος δεν κατάλαβε και ποτέ γιατί τα ίδια τα κόμματα κατέβαζαν 12 υποψηφίους ενώ γνώριζαν ότι από αυτούς δεν θα εκλεγούν παρά μόνο οι δύο-τρεις. Επαναλαμβάνω ότι η Εστονία, να διευκρινίσω εδώ, έχει έξι βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε ο κόσμος δεν καταλάβαινε τι νόημα έχει να περιμένει κανείς ότι θα πρέπει να ψηφίσει περισσότερους. Και σύν της άλλης είναι και εντελώς άγνωστες οι δραστηριότητες των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κόσμος στην Εστονία μιλάει για τη διαφθορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τους υψηλούς μισθούς, αλλά όχι για τις πολιτικές δραστηριότητες. Επίσης υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία προκαλούν το ενδιαφέρον των πολιτών όπως ας πούμε η κοινή γεωργική πολιτική και μόνο μέσα από πρακτικά παραδείγματα μπορεί το κοινό στην Εστονία να ενδιαφερθεί σαν παράδειγμα για την κοινή αλλιευτική πολιτική στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική μάλλον Θάλασσα αν είναι δυνατόν ε, ακριβώς η κοινή αλλιευτική πολιτική να βοηθήσει τους εσχολούμενους ε, με την αλληλεία, τότε θα υπάρξει και αύξηση του ενδιαφέροντος ε, των εσθονών στις ευρωεκλογέ. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την αλληλεία φυσικά, αλλά και για την απασχόληση, την πράσινη απασχόληση, σαν μέσο αύξησης της απασχόλησης γενικότερα τις συνέπειες ε, της ε, παινίας, μια ολόκληρη σειρά από θέματα τα οποία θα έλεγα παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Για τα μέσα ενημέρωσης ε, δεν ξέρω αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει κάποιες αλλαγές τον τελευταίο καιρό. Στην Εστονία κάθε Τετάρτη υπάρχουν συζητήσεις διακομματικές και οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων κάνουν εισαγωγή για διάφορα θέματα και τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σπάνια ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Μένει πολλά να γίνουν λοιπόν. Στην Εστονία θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει μια έλλειψη πολιτικής ευρωπαϊκής κουλτούρας και τα πολιτικά κόμματα ίσως σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουν πολλή δουλειά να κάνουν ακόμα. Θυμίζω ότι και οι κοινοβουλευτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να πιέσουν προς την κατεύθυνση αυτή σχετικά με την ηλικία για τη συμμετοχή στις εκλογές. Φυσικά και θα πρέπει να είναι ενιαίο σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, αν προτείνεται τα 16 χρόνια, αυτό ίσως να μην γίνει δεκτό στην Εστονία. Όπως επίσης δεν θα υποστηριχθεί και η κατώτερη ηλικία των 25 για την ε, ε, κάθοδο στον εκλογικό στίβο. Νομίζω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις πάντως είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για να βρεθεί μια λύση στο μέλλον. Οι δύο τελευταίοι αγορητές ε, μένουν ακόμα και μετά πρέπει να δώσω και λίγο χρόνο στον κύριο Ντάφ για να δώσει τις ενδεδειγμένες απαντήσεις. Δύο λεπτά λοιπόν το πολύ στους δύο τελευταίους ε, Τον Πορτογάλο κύριο Φελίπε και την συνάδελφο Μορβάη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Φιλίπε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για μια σειρά από τα ζητήματα της συζήτησης. Η Συζητήσει βέβαια αυτές δεν εκφράζουν το δικό μου κοινοβούλιο, είναι προσωπικές παρατηρήσεις γιατί δεν έχουμε κάνει κάποια τέτοια συζήτηση ακόμα. Να τονίσω ωστόσο ορισμένα πράγματα. Πρώτον, είναι όντως μια σημαντική συζήτηση που παρουσιάζει προφανώς ωστόσο σειρά δυσκολιών όπως προείπησε και από τι σημερινέ συζητήσει. Να τονίσω δύο πράγματα. Καταρχάς, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ναι μεν χρειάζεται να υπάρχει ενιαία εκλογική διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν σεβαστές και οι εκλογικές παραδόσεις των διαφόρων χωρών. Δεύτερον, να εκφράσω κάποια επιφυλακτικότητα για την ιδέα αυτού του πανευρωπαϊκού, της πανευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας ως εργαλείο ενίσχυσης της ταύτισης του Ευρωπαίου πολίτη με τις ευρωεκλογές. Ήδη αναφέρθηκε ότι οι ευρωεκλογές από πολλούς θεωρούνται στην πραγματικότητα εθνικές εκλογές και η ψήφος ε, εκφράζεται με βάση την εθνική κατάσταση ή ε, ε, επιβραβεύοντας ή μεμφόμενη την κυβέρνηση και όχι για την εκλογή ευρωβουλευτών αυτών καθευτών. Αυτό μειώνει την συμμετοχή, όπως το είδαμε άλλωστε μέχρι τώρα. Ωστόσο, αν δεν υπήρχε η εθνική διάσταση στις ευρωεκλογέ, η συμμετοχή θα ήταν ακόμα χαμηλότερη κατά την άποψή μου, διότι πάρα πολλοί ψηφοφόροι πηγαίνουν σε εκλογές αυτές μόνο και μόνο γιατί θεωρούν ότι είναι εθνικές δεν είμαι βέβαιος λοιπόν ότι η ενιαία εκλογική περιφέρεια θα κινητοποιήσει τους πολίτες περισσότερο. Η εγκύτητα των θεσμών με τον πολίτη σχετίζεται και με την γνώση του συγκεκριμένου υποψηφίου από τον ψηφοφόρο. Αντίθετο ωστόσο, πολλοί ψηφοφόροι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι οι αποφάσει τη Βρυξέλλε λαμβάνονται μακριά από του ίδιου. Άρα το ζήτημα είναι να καλύψουν το δημοκρατικό έλλειμμα εκεί. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που σας ε, διέκοψα. Να το πω αυτό και στην ε, συνάδελφο Μολβάη. Δύο λεπτά παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να λάβετε τα έγγραφα μπροστά σας. Πρόκειται για ένα παράρτημα, ε, για ένα κείμενο νομικής πράξης. Στη σελίδα 10 είναι στα Ουγγρικά και εκεί πρόκειται για τις ε, τροπολογίες. Έχουμε λοιπόν τις τροπολογίες για το κείμενο της ε, νομοθετικής πράξης και ήδη ε, στο πρώτο άρθρο έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Ε, αφορά την πράξη περιεκλογή του 1976. Σε κάθε κράτος μέλος λέει, μάλλον όχι, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται ως αντιπρόσωποι των πολιτών της με αναλογικό σύστημα. Στην ε, τροπολογία μιλάμε για αντιπροσώπους των πολιτών. Δηλαδή τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή αντιπρόσωποι τους ε, κατ' ουσίαν έχουν διαφορετική εντολή. Εγώ είμαι βουλευτής ε, του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να εκπροσωπώ τους πολίτες της Ουγγαρίας. Βλέποντας λοιπόν αυτή την ε, τροπολογία, κάτι τέτοιο μου απαγορεύεται, γιατί στην πρώτη τροπολογία αναφέρεται ότι εγώ πρέπει να εκπροσωπώ τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο πολίτη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο πολίτες της Ουγγαρίας. Ή παριθμόν, είναι η τροπολογία λέει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ψηφίζουν ονομαστικά και δεν δεσμεύονται. Ψηφίζουν ατομικώ και προσωπικώ. Δεν δεσμεύονται από οδηγίε, ούτε δέχονται δεσμευτική εντολή. Η τροπολογία λέει να διαγραφεί αυτό. Πρόκειται για την τροπολογία υπαριθμών 1 και την υπαριθμών 9. Αυτές μας ενδιαφέρουν. Ο εισηγητή με αυτέ τι δύο τροπολογίες σε τι αποσκοπεί και γιατί θέλετε να αλλάξετε την ε, εντολή ε, των, ε, που λαμβάνει ο Ευρωβουλευτής. Ο κύριος Νταφ έχει το λόγο. Αν έχει την καλοσύνη, όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Πρόεδρε, ευχαριστώ τους 26 συναδέλφους που συνέβαλαν στη συζήτηση. πίστευα και το προσδοκούσα ότι θα ήταν και εκτεταμένη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους ε, συναδέλφους να εκφράσουν τις αμφιβολίες τους για την ανάγκη μεταρρύθμισης. Αυτό είναι κατανοητό. Ελπίζω, ωστόσο, όπως είπαν και οι περισσότεροι, ότι οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν το ξεκίνημα μιας βαθύτερης ε, συζήτησης και μελέτης για την ενίσχυση της, νομικής, της λαϊκής νομιμοποίησης της το και αν κάποιοι δεν το θέλουν αυτό. Το σεβόμαστε. Ωστόσο, παρά το σεβασμό προς όσους ε, έχουν μια, ευρω, μια εθνικιστική προσέγγιση, τούτο δεν αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία. Δεν ζητάμε να αλλάξει τη συνθήκη. Η συνθήκη άλλαξε την περιγραφή της ε, λειτουργίας των μελών του Κοινοβουλίου ως εκπροσώπων των πολιτών της Ένωσης. Η συνθήκη το λέει αυτό και εγώ στις προτάσεις μου προσπαθώ να αντικατοπτρίσω την αλλαγή αυτή. Απαντώντας με πρακτικές προτάσεις υλοποίησης της αλλαγής αυτής. Προφανώς σε τέτοια εγχειρήματα πάντα υπάρχουν ε, Συνέπειε που δεν τι περίμενε κανείς. Δηλαδή οι προτάσει που στι Βρυξέλλε θεωρούνταν ε, ε, εύλογε να, να δημιουργούν προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να μελετήσουμε προσεκτικά το κείμενο. Για παράδειγμα, η πρόταση για την περιφερειοποίηση των εθνικών ε, εκλογικών περιφερειών στα μεγάλα κράτη της Ένωσης, καταλαβαίνω ότι στην Ισπανία δημιουργεί σοβαρά, σοβαρότατα ε, ζητήματα. Είναι όμως εξαιρετικά δημοφιλής στη Γαλλία. Οι Γερμανοί μπορεί να θεωρούν ότι αυτό είναι περιττή μεταρρύθμιση διότι ήδη διαθέτουν στο εσωτερικό του κράτους την ομοσπονδιακή τους δομή. Η πολιτική επιστήμη ωστόσο λέει ότι ο ψηφοφόρος χρειάζεται μία εκλογική περιφέρεια σε κατανοητή, διακριτή, σε κατανοητό και διακριτό μέγεθος, με το οποίο να μπορεί να ταυτιστεί. Μία εκλογική περιφέρεια στα όρια του κράτους δηλαδή μια εκλογική περιφέρεια που καλύπτει όλο το κράτος, απέχει πολύ από τον πολίτη. Δεν είναι σωστό αυτό που είπαν κάποιοι συνάδελφοι ότι οι ευρωβουλευτές είναι αναγνωρισμένοι στο εκλογικό πλαίσιο των χωρών τους. Υπάρχουν εξαιρέσεις. From the citizens... Οι περισσότεροι από εμά δεν βρισκόμαστε στο μυαλό των πολιτών μας όταν σκέφτονται την πολιτική καθημερινότητά τους. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σοβαρά το ζήτημα του μεγέθους των εκλογικών περιφερειών. Επίσης πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να προσπαθήσουμε να βγούμε από την αποκλειστικά εθνική νοοτροπία. υπάρχει μία αυξανόμενη ομάδα ψηφοφόρων που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως έχοντον πολλές ταυτότητες, εθνική, περιφερειακή και ευρωπαϊκή. Μπορούμε και που μπορούν απλά και μόνο να εκτιμήσουν την ιδέα ενός μιας μεταεθνικής δημοκρατίας. και που αναζητούν πολιτικά κόμματα τα οποία θα μπορέσουν να εκφράσουν πιστά τις δικές τους προσδοκίες. Ενώσο ο πολίτης δεν Μπορεί ο πολίτη να μην αναγνωρίζει το ότι η Ευρώπη μπορεί να απαντήσει στην, ε, στις προκλήσεις της ε, ε, παγκοσμιοποίησης, αλλά καταλαβαίνει ότι και τα εθνικά πολιτικά κόμματα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές, δεν δίνουν λύσεις στις πραγματικές ανάγκες. Δεν νομίζουν οι περισσότεροι πολίτες ότι τα οι ισχυρισμοί των, πολιτικών, των εθνικών πολιτικών κομμάτων ότι η, δημοκρατία η εθνική δημοκρατία λύνει όλα τα προβλήματα. Η αμφισβήτηση αυτής της έννοιας, της θέσης αυξάνεται. Υπάρχει όλο ένα και περισσότερο και περισσότερη επίγνωση της διεθνικής διάστασης των σημερινών σχέσεων εξουσίας. Τα γεγονότα είναι ότι εμπολής η εξουσία σήμερα έγκυται στις Βρυξέλλες και χρειάζεται μία ισχυρή αντιπροσωπευτική δημοκρατία που να μπορεί να ζητήσει από αυτή την εξουσία να λογοδοτεί. Θα ήταν λάθος να δεχθούμε ως ε, αμετάβλητη την υφιστάμενη κατάσταση. Νομίζω ότι η συζήτηση που έχουμε εδώ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και είναι κρίμα που η συζήτηση, οι συζητήσεις αυτές δεν εκφράζονται στις προεκλογικές εκστρατείες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις πολιτικές ομάδες διαμορφώνονται οι θέσεις. Να θυμίσω στην κυρία Μορβάη ότι μετέχουμε εμείς ως εθνικές αντιπροσωπείες σε πολιτικές ομάδες που δουλεύουν. Αυτό ωστόσο δεν αντικατοπτρίζεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εκλογ... της εκλογικής πολιτικής έξω από το Κοινοβούλιο, ούτε στον τύπο. Και πρέπει να σας πω ότι οι εκπρόσωποι των μέσων με παρότριναν να πιέζω, να, να προωθήσω αυτή την ιδέα της υπερεθνικής εκλογικής ε, περιφέρειας. Θεωρούν ότι πουλάει διαφημιστικά, ότι θα ήταν ενδιαφέρον να δουν τις ε, σημαντικές ε, συγκρούσεις προσωπικότητων από τις λίστες αυτές και τα ζητήματα, τα βασικά πολιτικά ζητήματα που θα θέτουν. Φερρυπίν, τα βασικά μεγάλα, τα μεγάλα σημερινά ερωτήματα, το μέλλον του νομίσματος, το μέγεθος, τα όρια της Ένωσης, τα ζητήματα μετανάστευσης. Οι πολύ σοβαρές, προβεβλημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και που θα μπορούν να αντιμετωπιστούν με ξεκάθαρο και που δεν μπορούν να, συγγνώμη, να αντιμετωπιστούν με ξεκάθαρο τρόπο στο υφιστάμενο εθνικό πλαίσιο. Πολλοί ομιλητέ εξέφρασαν ανησυχίε για το ενδεχόμενο να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των εθνικών πολιτικών κομμάτων. Το δέχομαι ότι θα υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός ανταγωνισμού από αυτή τη στιγμή. Και αυτό το θεωρώ ως κάτι καλό. Να παροτρύνουμε δηλαδή τον ανταγωνισμό σε επίπεδα των πολιτικών κομμάτων για μια δημοκρατία. Να τονίσω και πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος θα αντικατοπτρίσει τη βαθύτερη ενοποίηση που έχουμε διοικητικά και οικονομικά αλλά και στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο ισχυρισμό ότι ο κόσμος δεν θα παρακολουθήσει, δεν θα, καταλάβει τις προτάσεις που κάνω. Υποστηρίζω απόλυτα την αμφισβήτηση της άποψης αυτής από τον Τζον Τζολάινεν, ότι δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις δεν πάνε αρκετά μακριά για να αλλάξουν επαναστατικά την ευρωπαϊκή πολιτική. Προφανώ δεν μπορεί να κάνουμε τεράστια άλματα, αλλά από την άλλη μεριά προχωράμε αρκετά για να αλλάξουμε, να μετατρέψουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα της επόμενης ε, προεκλογική καμπάνια. Μου είπανε γιατί 25 σε αυτή τη λίστα. Για πρακτικούς λόγους. 25 ονόματα μπορούν να βγουν σε ένα ψηφοδέλτιο τέλο πάντων που δεν θα είναι τεράστιο. Και ένα βασικό στοιχείο οποιασδήποτε εκλογική μεταρρύθμιση είναι, είναι πρακτική. Για προφανείς λόγους Πιστεύω ότι ήταν λάθος να πούμε 27 υποψήφοι. Γιατί αν συνέβαινε αυτό και μπαίνει η κρατή μετά και γινόμασταν 28, θα έλεγε ο κόσμος ότι κάθε κράτος θα μπορεί να βάλει στη λίστα αυτή ένα έξτρα μέλος. Που δεν είναι σωστό. θα μπορούσε να είναι σωστό τυχαία από μια δημοκρατική τύχη. Αλλά δεν είναι αυτή η πρόθεση της πρότασης που είναι να σπάσει η σχέση ανάμεσα στο κράτος και την ηθαγένεια από τη μια μεριά και τη σύνθεση του Κοινοβουλίου από την άλλη. Πολλοί ρώτησαν γιατί προτείνω να συμπληρώσουμε, να προσθέσουμε τους βουλευτές αυτές και όχι να τους ε, ξηρίσουμε από τα, κράτη, από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Πολιτικά ωστόσο θα έλεγα αν αρχίσουμε να ζητούμε από τα κράτη να δεχτούν μείωση του αριθμού των εθνικών σε εισαγωγικά βουλευτών δεν θα τους αρέσει πολύ. Κάποιοι κατέκριναν το ότι το κοινοβούλιο θα γινόταν πολύ μεγάλο. Πρέπει να πω ότι διαφωνώ. Το κοινοβούλιο δουλεύει αυτή τη στιγμή εξαιρετικά σκληρά όσο προχωρά ταχύτερα ο ρυθμός ενοποίησης. Έχουμε εξαιρετικά καλή υποστήριξη, θα έχουμε εξαιρετικά καλή υποστήριξη από την παρουσία εδώ ε, μεγάλων ευρωπαϊκών προσωπικότητων. Τώρα, για το ερώτημα, θα υπάρχουν δύο κατηγορίες βουλευτών. Η απάντηση είναι ναι, προφανώς. Αλλά και τώρα υπάρχουν διάφορες κατηγορίες βουλευτών που δουλεύουν και ασκούν το λειτουργήμά τους με διαφορετικό τρόπο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι μπορούσα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ ωστόσο ιδιαίτερα για την εξαιρετικά πλούσια συμβολή στην περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου που θα έχουμε στο Κοινοβούλιο και στις Εθνικές Πρωτεύουσες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς ε, κύριε Νταφ. Ε, πριν λοιπόν ε, κλείσουμε και ολοκληρώσουμε την πρωινή μας συνεδρίαση, θα ήθελα να δώσω λόγο στην κυρία Γκουρμάη, την Αντιπρόεδρο, για να πει και αυτή δύο λόγια, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πια χρόνο, γι' αυτό και εγώ θα μιλήσω πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνάντηση. Εγώ είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι πρέπει να συναντιόμαστε συχνότερα με τους ε, εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πρέπει να συζητάμε τα μεγάλα θέματα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι θα συνεχίσουμε τη συνάντησή μας ε, και σήμερα το απόγευμα θα μιλήσουμε για την πρωτοβουλία των πολιτών. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερα ευρωπαϊκά θέματα. Ε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Νταφ, ο οποίος προσφέρθηκε να συντάξει αυτήν την έκθεση. Το νομοσχέδιο αυτό, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ε, είναι πολύ παλιά. Πρέπει να προετοιμαστούμε στα καινούργια δεδομένα. Και υπάρχουν πολλά θέματα όπου πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι από το 1979 ε, μειώνεται φθήνη συστηματικά τον ενδιαφέρον για την Ευρώπη. Στις τελευταίες εκλογές μόνο το 46% των πολιτών συμμετείχαν σε εκλογές. Άρα δηλαδή οι σχέσεις τους με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν είναι πολύ καλές. Και σήμερα το απόγευμα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε μικρά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Εξάλλου είμαι πεπισμένη το ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει αυτό να αναφερθεί στην έκθεση, ότι πρέπει στο Κοινοβουλίο να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες. Εντάξει, έχει αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά χρειαζόμαστε και άλλες. Ευχαριστούμε κύριε Νταφ, ευχαριστούμε πρόεδρε και ελπίζω να συναντηθούμε σήμερα το απόγευμα και να μιλήσουμε για την πρωτοβουλία των ε, πολιτών. Ε, πολύ ωραία, στις 3 ε, και θα ξανασυναντηθούμε και νομίζω έχουν μοιραστεί οι, προσκλήσει οι προσκλήσεις ε, για το μεσημεριανό γεύμα. Πολύ γρήγορα, το άρθρο 12 το γνωρίζετε. Λέει, τα, Ευρω... κοινοβούλια, τα εθνικά ε, συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ένα τρίτο κοινοβουλίο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προφανώς ε, διεκδικεί τη δική του την αυτονομία. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν δικό τους ρόλο, κάνουν δική τους δουλειά, που είναι κυρίως ο έλεγχος των εθνικών κυβερνήσεων. Όμως, όσον αφορά στη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το άρθρο 23 αποδίδει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αρμοδιότητα να επεξεργαστεί μεταρρύθμιση για να υπάρξει νέο εκλογικό σύστημα. Μετά το δεύτερο κόμμα όμως λέει ε, προφανώς το κείμενο αυτό πρέπει να εγκριθεί και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Άρα δηλαδή αυτή η συνεδρίαση μπορεί να είναι μόνο το εναρκτήριο λάκτισμα και εγώ πιστεύω ότι κάτι το ε, θεσμικό, η Κόζακα ας πούμε, εκεί είναι ο σωστός χώρος για να συνεχιστεί όλη αυτή η προβληματική. Γιατί όπως υπόθηκε το θέμα είναι στρατηγική σημασίας, αφορά το σύνολο της Ευρώπης δεν είναι κάτι το τεχνητό. Νομίζω ε, ότι είναι κάτι το ρεαλιστικό, το ε, σημαντικό, αρκεί να σκεφτούμε ότι ένας πόλεμος μεταξύ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο δεν έλαβε χώρα, αλλά ούτε καν μπορεί να μπει στην, ε, στο χώρο του εφικτού. Άρα δηλαδή δεν είναι ανέφικτο αυτό το οποίο συζητάμε. Δεν είναι δευτερεύουσα σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή σας όρεξη.